So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στο τρίτο πάνελ ε, αυτής της διακοινοβουλευτικής ε, διάσκεψης. Ε, καλωσορίζω θερμά και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημερινά θέματα της απογευματινής συζήτησης θα είναι στο πρώτο τμήμα τι είναι η κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού αλφα Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών καθορισμού μισθολογίων και στο δεύτερο τμήμα από τις 4.30 και μετά θα ασχοληθούμε με τις επενδυτικές πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, επενδυτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτικής ανάπτυξης δεξιοτήτων. θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τα Εθνικά Κοινοβούλια που απάντησαν μετά από πρότασή μας και Δέκα συνολικά απαντήσεις έχουν φτάσει στα χέρια μας. Και πριν πω στην ημέρηση αδιάταξη θέλω να καλωσορίσω θερμά το Ζωζ Έγγελ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Ασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, Σάμπρ Ντεπιτέ. Και περιμένουμε ακόμα τον κύριο Νίκο Μανιό, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Βουλής των Ελλήνων δηλαδή είναι στο Κοινοβούλιο και ξέρω ότι είναι καθοδόν. Στους διαδρόμους μάλλον τον έχουν ε, καθυστερήσει κάποιε συζητήσει ή κάποιες συνεντεύξει. Πριν μπούμε στη συζήτηση θα ήθελα να θυμίσω ότι ε, θέλουμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με το πρωί ε, και θα σας παρακαλούσαμε αν θέλετε το λόγο να συμπληρώσετε κάποια ε, φύλλα που έχετε κάτι σελίδες. Υπάρχει η λευκή σελίδα για το πρώτο τμήμα της συζήτησης για το τριπλό α και ένα κίτρινο χαρτί που θέλετε ε, να συμπληρώσετε αν θέλετε να μιλήσετε ε, στο δεύτερο πάνελ για να μπορέσουμε να τα μοιράσουμε. Και παρακαλώ να είναι βανάγνωστα γιατί σήμερα το πρωί οι συνάδελφοι είχαν κάπως ιατρικό γραφικό χαρακτήρα και δεν μπορούσαμε κάθε φορά να μαντεύουμε τα ονόματα. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Θα ε, προσπαθήσουμε λοιπόν έτσι να δώσουμε και το λόγο σε όλους όσοι τον ζήτησαν. Οπότε να πούμε περιορισμός δίλεπτο για κάποιους συναδέλφους. Ε, αυτό είναι έκπληξη, αλλά οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν έχουν δύο λεπτά χρόνο ο, Αγόρευση ε, πανηγυρίζουν. Ήρθε ο κύριο Μανιό, καλώ ορίσατε κύριε Μανιέ. Οι περισσότεροι λοιπόν ε, ε, οι βουλευτές είναι συνηθισμένοι οι ευρωβουλευτές να έχουν δύο λεπτά χρόνο αγόρευση. και ξέρω ότι πολλές φορές τα Εθνικά Κοινοβούλια έχετε περισσότερο χρόνο αγόρευση και σας ζηλεύουμε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα κάνουμε με το χρόνο και θα παρεμβαίνω όταν κάποιο μακρηγορεί και σας παρακαλώ να με συμπαθάτε. Αυτό που θέλω είναι να μιλήσουν όλοι, όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, μια μικρή εισαγωγή. Τι είναι η κοινωνική βαθμολόγηση τυπρού ΑΛΦΑ. Ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ το πρότεινε αυτό ήδη από το 2014 σε μια ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το όλο κατέληξε σε μια συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικού δικαίου τον Οκτώβριο του 2015 συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια συζήτηση ανατολισμού συνεννοήθηκε για το θέμα αυτό και βολιδοσκόπησε την κατάσταση και το έχει εντάξει και στο πρόγραμμα εργασίας για το 2016. Έκτοτε από το Γενάρη του 2016 συμπληρώθηκε και με άλλους τομείς και συγκεκριμενοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασε από το στάδιο της βολιδοσκόπησης και άρχισαν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με αιρετούς αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Για να καταλήξουμε σε ένα ενδεχόμενο κοινωνικό πυλώνα ε, για τα κοινωνικά δικαιώματα και εμείς στην Επιτροπή ε, Απασχόλησης πιέζουμε πάρα πολύ να γίνει ευρεία συζήτηση, διαβούλευση. Στο μεταξύ άρχισαν να συγκεκριμενοποιούνται κάποια θέματα, κάποιες επικεφαλίδες ας πούμε ενός τέτοιου κεφαλαίου. Παράδειγμα, νέα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στον 21ο αιώνα. Επίσης πρόκειται για το θέμα της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας που πρέπει να καταπολεμηθούν και κοινωνικά δικαιώματα, ισορροπία ε, εργασιακού και ιδιωτικού βίου για εργαζόμενους γονείς. Έχουμε μια ευρωπαϊκή ατζέντα, ένα θεματολόγιο για προσόντα και δεξιότητες και το πακέτο της κινητικότητας των εργαζομένων. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό και πιέζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες ε, θα κάνει κάποιες προτάσεις και αν θέλουμε να δούμε ποια τα κοινωνικά δικαιώματα, οι ελάχιστες προδιαγραφές, είναι πάρα πολλοί ορισμοί που θα βρείτε ε, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και σε ε, διάφορες συμβάσεις ε, του Διεθνού Οργανισμού Εργασίας. Το θέμα είναι τώρα να γίνουν όλα αυτά πια πιο χειροπιαστά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο ευρωζώνης και να κληθούν όλες οι υπόλοιπες χώρες να συνεργαστούν σε αυτό το θέμα. Προετοιμάζοντας λοιπόν τη σημερινή μας συνεδρίαση, κάναμε ένα ερωτηματολόγιο που σας στείλαμε. Δεν θέλω να σας επαναλάβω τις ερωτήσεις, τις έχετε άλλωστε ε, οι απαντήσεις που λάβαμε θα συμπεριληφθούν στη σημερινή συζήτηση και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει στις ερωτήσεις μας είναι και το εξής. Οι κοινωνικοί εταίροι πώς μπορούν σε εθνικό επίπεδο πια να συμμετέχουν σε μια τέτοια συζήτηση. Επίσης τίθεται το θέμα των, ε, των Συμβουλίων Ανταγωνισμού ένας μηχανισμός ορισμού των μισθών. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίμαχο και σήμερα θα πρέπει να μας απασχολήσει η σχέση με αυτό που ζητάει ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ, ίση αμοιβή για ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας ε, και χώρο δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ θετικό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν αυτά να μεταφραστούν σε νομοθεσία προς το παρόν ακόμα δεν είναι λυμένο. Αυτά τα εισαγωγικά για να σας ε, εισαγάγω στο θέμα. Ελπίζω να μην ε, κάλυψα πάρα πολύ ε, αυτά που θέλουν να πούν οι δύο μιλητές μας. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον Ζωζέγγελ και μετά στον Νίκο Τομανιό. Μανιό. μετά θα μπούμε στη συζήτηση. Παρακαλώ. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος Επιτροπής Εργασίας Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλή των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Χέντελ, ο οποίος μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για ένα ζήτημα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι εδώ και πάνω από 50 χρόνια ορισμένες χώρες, εκ των οποίων και το Λουξεμβούργο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας χώρος σταθερότητας και ειρήνης, τον οποίο θεωρούσαμε πάρα πολύ δεδομένο για πάρα πολλά χρόνια και που δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί χωρίς την πρώτη αυτή συμβολή των πρώτων αυτών κρατών. Το 1950 οι υπογράφοντες στη διακήρυξη Σούμαν είχαν θέσει ως στόχο να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας αυξανόμενης πρόοδου και θεωρώ ότι ε, ο στόχος αυτός ήταν ιδιαίτερα δικαιολογημένο. Οι υπόλοιπε συνθήκες δώσανε νέα όθηση σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό κοινωνικό όραμα το οποίο για πάρα πολύ καιρό είχαμε λησμονήσει. Η συνθήκη της Λισαβόνας τόνωσε την πρόθεση της απασχόλησης, την ε, διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα αυτά θεωρούνται πλέον στο επίκεντρο του κοινωνικού ευρωπαϊκού οράματο. Αυτή τη στιγμή όμω βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικότατα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή από το γεγονό ότι έχουμε ιστορικά επίπεδα ανεργία, ένα τεράστιο χάσμα ανισοτήτων, ένα τεράστιο επίπεδο φτώχεια και ένδυα που πλήττει του Ευρωπαίου πολίτε. Και βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερο χάσμα που χωρίζει πλέον τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργία των νέων, καθώς επίσης και η φτώχεια και η ένδια που πλήττει τα παιδιά, καταδεικνύουν ότι πραγματικά θα πρέπει να επικεντρώσουμε εκ νέου το ευρωπαϊκό εγχείρημα στην κοινωνική του διάσταση, αν πραγματικά θέλουμε να αποφύγουμε μια κοινωνική διάσπαση, καθώς επίσης και μια αδιαφορία ή ακόμα και αντίθεση των Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και θέλουμε να αποφύγουμε επίσης την άνοδο του εξτρεμισμού και του λαϊκισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονός ότι μολονότι υπάρχουν ε, κοινωνικές και οικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες αποτελούν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν απειλή και για την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για αυτό το λόγο να τονώσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια διάσταση που πολλές φορές είχαμε παραβλέψει, ή στιγματίσει πάρα πολλές φορές και είχαμε προωθήσει περισσότερο την οικονομική και νομισματική σύγκληση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεντρωμένη εκ νέου στους Ευρωπαίους πολίτες, αυτή πρέπει να είναι η βάση της νέας συνεργασίας των κρατών μελών της Ένωσης. Αυτή η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να προβλέπει την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια καλύτερη βάση για την απασχόληση, την εργασία, τις συνθήκες απασχόλησης και θα πρέπει να θέτει ως στόχο την καταπολέμηση του φορολογικού, μισθολογικού ντάμπινγκ και του κοινωνικού αποκλεισμού προωθώντας παράλληλα το κοινωνικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε μια ισχυρή κοινωνική προστασία, σε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας το οποίο θα βασίζεται με τη σειρά του στον κοινωνικό διάλογο. Η κοινωνική λοιπόν διάσταση της Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλε μα τι πολιτικές, είτε αυτέ είναι οικονομικέ είτε είναι χρηματοπιστωτικέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνική αυτή διάσταση να τεθεί στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μα ιδίω στα επόμενα βήματα τη ολοκλήρωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση μπορεί να προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο προκειμένου να προωθήσει με τρόπο ισορροπημένο μια πιο ισχυρή ανταγωνιστικότητα, μια καλύτερη διαφορετική σύγκληση, καθώς επίσης όμως και μια πολιτική ένταξης όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κοινωνικές λοιπόν αυτέ πολιτικές και η πολιτική απασχόληση θα πρέπει να συντονιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο λαμβάνοντα υπόψη τις ιδιαιτερότητέ τους. Αν πραγματικά επιθυμούμε να προωθήσουμε μία πιο κοινωνική Ευρώπη, τότε πραγματικά θα πρέπει να καταλήξουμε και σε μία κοινωνική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ακριβώς αυτή η κοινωνική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χωρίς την πολιτική αυτή δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το κοινωνικό αυτό ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται βέβαια και από μια μεταρρύθμιση των ε, κοινωνικών μας μοντέλων και των ε, μοντέλων κοινωνικής πρόνοιας. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, το Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια της ε, προηγούμενης προεδρίας του, αποφάσισε να θέσει τον Ευρωπαίο πολίτη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αποφασίσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτέλεσε σημαντικότητα προτεραιότητα και της κοινοβουλευτική διάστασης της Λίξεμβουργιανής προεδρία. Και για αυτό το λόγο διοργανώσαμε τρει διακοινοβουλευτικέ ε, συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας και μάλιστα τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε και μια τέτοια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση των βουλευτών των Επιτροπών Απασχόλησης Ευρωπαϊκή Ένωσης. Προσπαθήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να δούμε πώς θα δώσουμε νέο κοινωνικό πρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτό το περίφημο κοινωνικό τριπλό α. Θελήσαμε επίσης στα πλαίσια της Προεδρίας μας να περάσουμε από αυτό το κοινωνικό χάσμα, το κοινωνικό έλλειμμα, σε αυτό το κοινωνικό τριπλό α, σε επίπεδο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταβάλλουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μία οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, προκειμένου να ενισχύσουμε και το σχέδιο Juncker και να οδηγηθούμε σε μια νέα οικονομική ανάκαμψη και σε μια ισχυρή ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν απαραίτητε κοινωνικέ επενδύσει και όλο ιδιαίτερο θα πρέπει να γίνουν επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε μια ισοπαίδωση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα έρθουμε πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θα πάψουν πλέον να βλέπουν την οικονομική ολοκλήρωση και το ευρώ ως απειλή. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε σφαιρικά το κοινωνικό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να απεφύγουμε όλους αυτούς τους κινδύνους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής μας αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό να, τον, να τονίσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές πτυχές της οικονομικής μας πολιτικής. Υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι οι λύσει θα είναι εύκολε, αλλά παρόλα αυτά δεν προτείνουν τίποτα το ουσιαστικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε γι' αυτό ακριβώ το λόγο πιο φιλόδοξοι. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική σύγκληση προ τα πάνω. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μα όσον αφορά τα συστήματα κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε μια κοινωνική διάσπαση, μια κοινωνική διάλυση που θα είναι πραγματικά καταστροφική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως φοβούνται ορισμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια κοινά κοινωνικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στις απαραίτητες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε, όπω σα είπα, κοινωνικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερο συντονισμό λοιπόν των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συντονισμένα συστήματα μεταφορά των δικαιωμάτων συνταξιοδότηση από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερη αναγνώριση επίση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να βρούμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα μπορούσε να συνδυάσει μακροοικονομική ισορροπία και πάταξη της ανεργίας. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές. Ο αρμόδιος Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικών και κοινωνική ασφάλισης στην Ευρωπαϊ... στο Λουξεμβούργο έχει ακριβώ δώσει μάχη για τα ζητήματα αυτά και θεωρώ ότι και εμείς ως βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και ω μέλη των αντίστοιχων επιτροπών στα Εθνικά μα Κοινοβούλια θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ σημαντικέ προσπάθειε, οι οποίε θα πρέπει να περάσουν πρώτα από έναν ενισχυμένο διάλογο και από μια στενή συνεργασία μεταξύ ημών και μεταξύ των ε, κοινωνικών εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην ξεχνάμε όμω και τι χώρε εκείνε οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Όλοι από κοινού, τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις. Η οικονομική πρόοδο, ας μην το ξεχνάμε, συνάδει και συνδέεται με την κοινωνική πρόοδο. Τέσσερα στοιχεία κατ' είναι πολύ σημαντικά για μια κοινωνική Ευρώπη. Πρώτον, ανάπτυξη των κοινωνικών κοινών προτύπων. Δεύτερον, να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινωνική διακυβέρνηση, κοινωνικο-οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, προώθηση τη απασχόληση και τη κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Και τέταρτον, να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε επί ενό συγκεκριμένου θεματολογίου όσον αφορά τι κοινωνικέ επενδύσει. Μπορώ να επανέλθω αργότερα αν θέλετε στα σημεία αυτά. Κυρίες και κύριοι, από κοινού θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου η Ευρώπη να δώσει νέα πνοή στην κοινωνική της διάσταση. Από κοινού όλοι μαζί θα πρέπει να καταλήξουμε σε αυτή την κοινωνική βαθμολόγηση τριπλού α και θα πρέπει να προσαρμόσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο. Ας έχουμε λοιπόν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή σε μια εποχή που βλέπουμε ότι υπάρχει ρίζοσπαστικοποίηση και η αναδίπλωση στα κράτη-μέλη. Προφανώς δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να αναλάβουμε δράση. Το οφείλουμε αυτό στους πολίτες μας. Ας επικεντρωθούμε εκ νέου στα ουσιαστικά ζητήματα. Ας επικεντρωθούμε στα ζητήματα τα οποία μας ενώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Και πρόκειται για υποσχέσεις που από κοινού θα πρέπει να τηρήσουμε. Και μόνο μέσω της ελεγγύης μπορούμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να γεφυρώσουμε τις ανισότητες. Και είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών εκείνων οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός πραγματικού κοινωνικού συμφώνου. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζορ για την εισαγωγή. Η συζήτηση θα ακολουθήσει αφού ακούσουμε και τον Νίκο Μανιό, ε, τη δική του τοποθέτηση και παρουσίαση, γιατί ήδη ε, τροφή για συζήτηση έχουμε. Παρακαλώ, Νίκο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δίνετε διαμέσω εμού να εκφραστεί το ελληνικό ε, κοινοβούλιο. Ε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την πλευρά μας χαιρετίζουμε την προσπάθεια για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και δεσμευόμαστε πως το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα είναι ενεργό σε κάθε βήμα, κάθε προσπάθειες που θα ενισχύει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, όπως το ξέραμε. Ένα μοντέλο κοινωνικής προστασίας και δίκαιης κοινωνικής ανάπτυξης. Συζητάμε εδώ όμως μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και του ευρωπαϊκού εξαμήνου ένα πλαίσιο που κατά τη γνώμη μου αποκρισταλώνει τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικές οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί τουλάχιστον στη χώρα μου με βάση τα οικονομικά δεδομένα και τους κοινωνικούς δείκτες δεν οδηγούν στη βελτίωση των δημοσιονομικών. Δεν δημιουργούν άμεσες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και γενικότερα δεν ευνοούν τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των πολιτών. Πρόκειται για ένα πλαίσιο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι προωθεί τη σφιχτή δημοσιονομική προσαρμογή και όχι την κοινωνική δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά η Ελλάδα όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τη συμφωνία που έχει υπογράψει με τους θεσμούς επιχειρεί να διαχειριστεί τις πολιτικές αυτές και να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώντας όσο περισσότερο μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυ κοινωνικής προστασίας ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού. Τα σημεία που θεωρούμε σημαντικό να αναδειχτούν ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης είναι τα εξής. Πρώτον, η διαχείριση κρίσεων έχει επικεντρωθεί μέχρι τώρα στη δημοσιονομική εξυγίανση και στις μακροοικονομικές πτυχές με βασικό εργαλείο τη λιτότητα. Βλέποντας όμως τις κοινωνικές συνέπειες οφείλουμε να βρούμε άλλα εργαλεία ανάπτυξης και αντιμετώπισης των κρίσεων όπου η αξιοπρεπής και σταθερή απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές θα είναι στο επίκεντρο. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα πρέπει να στοχεύσουμε όλοι μαζί στο να ενσωματωθούν τα κοινωνικά κριτήρια σε όλους τους σχετικούς τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Δεύτερον, κάθε οικονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικές επιπτώσεις από την άσκησή της και να επικεντρώνεται στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Τρίτον, η κοινωνική βιωσιμότητα θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη χρειαζόμαστε εκ νέου ισορροπία με τη συμβολή των Υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ενισχυμένη συνεργασία και καλύτερη συνέργεια ιδιαίτερα μεταξύ του Συμβολίου Απασχόλησης και της Κοινωνικής πολιτικής και καταναλωτών. Και επίσης συνεργασία και με το Συμβούλιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, το γνωστό ΕΚΟΦΗΝ. Τέταρτο, θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, ακόμη και στο καθώς και την ενεργό συμμετοχή και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέμπτον, οποιαδήποτε πολιτική για να είναι οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και επομένως να απαντά στα προβλήματα με ικανοτικό τρόπο πρέπει να διασφαλίζει την εξισορρόπηση των δύο διαστάσεων της κοινωνικής και της οικονομικής. Ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων επισημαίνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει νομοθεσία που προωθεί τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, συχνά όμως είτε δεν εφαρμόζεται είτε δεν είναι αρκετή. Αυτό που χρειάζεται είναι δημιουργία μιας διαδικασίας σύγκλησης προς τα πάνω τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και εντός των κοινωνιών έχοντας στον πυρήνα, στον πυρήνα της τη λογική της δημιουργίας θέσεων αξιοπρεπούς και σταθερής εργασίας, τη διαφύλαξη και προώθηση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, την προστασία και τον εμπλουτισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις μεταβαλλόμενες συνθήκες των κοινωνιών της Ευρώπης και του κόσμου της εργασίας. Θα πρέπει να χρησιμεύει ως πηξίδα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δικαιοσύνης. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα πρέπει να προωθεί και να συμπληρώνει κάθε προσπάθεια για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν θα επιτελεί πραγματικά το ρόλο του. Θα έχει ένα όνομα που θα είναι κενό περιεχομένου. Φυσικά οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις των πολιτών θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας. Από την αρχή κάθε διαβούλευση μέχρι την τελική εφαρμογή και τη συνεχόμενη διαδικασία ελέγχου αξιολόγησης. Ειδική μνήμα θέλω να κάνω εδώ στο θέμα της συλλογική συνεννόησης των μισθών και της σημασίας. Και αυτό όχι μόνο γιατί το θέμα είναι στον τίτλο της σημερινή μας συζήτησης. Όλες και όλοι εδώ γνωρίζουμε τους δίκαιους αγώνες που έχουν δοθεί τους τελευταίους αιώνες στην Ήπειρό μας αλλά και αλλού στον κόσμο για να καθερωθεί το δικαίωμα στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις. Είχαμε καταφέρει ως Ευρώπη αυτό το δικαίωμα να θεωρείται ως βασικό και αυτονόητο. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν ισχύει αυτό για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει λοιπόν ισοτιμία και ισονομία ανάμεσα σε όλους τους εργαζόμενους της Ένωσης. Το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει καταργηθεί εδώ και κάποια χρόνια στη χώρα μου μέσα από τις πιέσεις της Τρόικα ακόμα και παρά τη σκληρή μάχη που εξακολουθεί να δίνει η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει αποκατασταθεί λόγω της στεναρής αντίθεσης των θεσμών. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων είναι όμως μια βασική δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό και πιστεύω πως θα πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες. Ως μέλη όλοι μας επιτροπών απασχόλησης στα κράτη μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουμε πως η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πρέπει, και πρέπει να παλέψουμε ώστε να υπάρχει ενιαία πανευρωπαϊκή δεσμευτική πρόβλεψη για την κατοχήρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της συλλογικής απόφασης των μισθών με το κράτος να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για τη στήριξη των εργαζομένων. Δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων με τέτοιου είδους παραλήψεις ή με δυνατότητα εξαιρέσεων κρατών μελών από την εφαρμογή τους. Πιο συγκεκριμένα τώρα, σύμφωνα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει σε δύο συμπληρωματικούς άξονες. Πρώτον, τον εξυγχρονισμό και την αντιμετώπιση των κενών της ισχύουσας νομοθεσίας για την κοινωνική πολιτική ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σημερινό εργασιακό περιβάλλον και να διασφαλίζεται ότι τα νέα μοντέλα εργασίας διατηρούν σωστή ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Εδώ οφείλουμε να προσθέσουμε ως Εθνικά και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως δεν μπορούμε να τηρούμε μια στάση ίσων αποστάσεων. Οι εργαζόμενοι είναι σαφώς ο πιο αδύναμος κρίκος αυτής της εξίσωσης και οποιαδήποτε πολιτική θέλουμε πραγματικά να είναι δίκαιη οφείλει να μεροληπτεί υπέρ των εργαζομένων. Δεύτερον, τον προσδιορισμό κοινωνικών συστημάτων βαθμολόγησης ιδίως όσον αφορά την έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια που, βασίζε, που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Και πάλι εδώ ως κοινοβούλια οφείλουμε να πούμε πως ειδικά σε αυτόν τον τομέα υποστηρίζουμε στεναρά την έννοια της σταθερής και ασφαλούς εργασίας και πως ιδιαίτερο ρόλο σε κάθε στάδιο μιας τέτοιας διαδικασίας θα πρέπει να έχουν οι ενώσεις και τα συνδικάτα των εργαζομένων βασικός σκοπός των όποιων κοινωνικών συστημάτων αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η εθνική και ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή, η αποφυγή κάθε είδους κοινωνικού ντάμπινγκ και η ανωδική σύγκληση όσον αφορά την ένομη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων. Αναφορικά με τον προσδιορισμό των κοινωνικών κριτηρίων ως παραδείγμα της αναφέρω πως θα μπορούσαμε να έχουμε τους δείκτες ανεργίας, το μορφωτικό επίπεδο, τη διαθεσιμότητα της φροντίδας των παιδιών, τη φορολογική επιβάρηση της εργασίας, μιας και έχουν αποδειχθεί ότι σχετίζονται με τα επίπεδα της απασχόλησης. Φυσικά, ο όποιος προσδιορισμός θα πρέπει να γίνει από κοινού μεταξύ των πολιτικών φορέων με ενεργή συμμετοχή των ενώσεων των εργαζομένων. Τελειώνοντας να πω ότι από όσο γνωρίζω το θέμα εδώ έχει συζητηθεί και στην Επιτροπή Απασχόλησης που συμβουλεύει σχετικά το Συμβούλιο και μας βρίσκει σύμφωνους ως εξής, στην εξής θέση. Οι προτάσεις που καταγράφονται για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων φαίνονται να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να μελετηθούν οι επιπτώσεις που έχουν προκύψει ήδη από την αλλαγή των σχέσεων εργασίας και από τις εφαρμοσμένες οικονομικές πολιτικές. Η επιμονή σε περιοριστικές πολιτικές που έχουν στόχο τη δημοσιονομική προσαρμογή με τα μέχρι τώρα αποτελέσματά τους αποδεικνύονται, αποδεικνύονται ότι κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τους στόχους των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές θα είναι χρήσιμες και θα φανούν ωφέλιμες αν διασφαλίζουν το δικαίωμα της υγείας, της παιδείας, της εργασίας και κατοικίας στους πολίτες κάθε κράτους μέλους. Εδώ επιτρέψτε μου να προσθέσω πως ειδική σημασία θα πρέπει να δοθεί σε στόχους που ενισχύουν τα παιδιά, τους νέους, τις εργαζόμενες μητέρες και τους ηλικιωμένους με συγκεκριμένα εφαρμόσιμα και χρηματοδοτούμενα μέτρα και όχι απλώς με υποδείξεις και αναλύσεις μιας και είναι οι πρώτοι που βάλλονται σε περιόδους κρίσης. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως τα κοινωνικά δικαιώματα είναι πανανθρώπινα και μας αφορούν όλες και όλους. Δεν θα υπάρξει πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αν δεν είναι συνολικός, αν δεν, δεν αφορά και δεν εφαρμόζεται για όλες και όλους όσους ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως της υπηκότητάς μας, της καταγωγής μας, του φίλου μας και του σεξουαλικού μας προσανατολισμού, των θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω στην καλή συνεργασία όλων μας και ότι δεν καταχράστηκα τον χρόνο. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Όταν καλούμε ομιλητές, πάντα τους ε, δίνουμε μια σύσταση για το πόσο χρόνο ομιλιά έχουν, αλλά αυτά που είπες εσύ ε, μας έδωσε πάλι τροφή προς συζήτηση και καθόλου δεν καταχράστηκε στον χρόνο, όχι. Λοιπόν, ε, ανοίγει συζήτηση, 12 συνάδελφοι ζητούν το λόγο και νομίζω ότι μπορούμε προς το παρόν να ορίσουμε ένα δίλεπτο χρόνο αγόρευσης για να προχωρήσουμε. Ο Ρόμαλς Ράτσοξ πρώτος από τη Λετωνία. Παρακαλώ. Parliament and European Social Rights. Ε, όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνέχισης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο της Λετωνίας και θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων επιλέξαμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που να επικεντρώνεται όχι μόνο στην ε, οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη και έτσι έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί ε, διακυβέρνησης ε, που παρέχουν μια ευρύτερη προοπτική σε κοινωνικά θέματα και ε, ενθαρρύνουν την ανταλλαγή απόψεων και το να εστιάζονται οι πόροι ώστε να αποφεύγεται ο κοινωνικός αποκλεισμός. Όσον αφορά το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα, η Λετωνία είναι μάλλον ε, επιφυλακτική. Φυσικά θα μπορούσε ε, να ωφελήσει σε κάποιους τομείς, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όσον αφορά την απασχόληση και την ε, κοινωνική πολιτική υπάρχουν ήδη μηχανισμοί σε εθνικό επίπεδο. Ο καθορισμός οι μηχανισμοί καθορισμού των μισθών επίσης πιστεύουμε ότι αποτελεί θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Στην ε, Λετωνία έχουμε αναθέσει το θέμα αυτό στους κοινωνικούς εταίρους ε, και ενώ σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή ε, την διαφορά. Επίσης έχουμε ένα τριμερές συμβούλιο που στόχο έχει να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση της οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τα συμφέροντα της κοινωνίας ε, και του κράτους ε, και να έχουμε στρατηγικά προγράμματα ε, πάνω σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα για να εγγυηθούμε την κοινωνική σταθερότητα και να αυξήσουμε την ευημερία σε όλη τη χώρα, καθώς και να αυξήσουμε την ευθύνη των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται και την εφαρμογή τους. Το Συμβούλιο ε, επίσης εξετάζει τις ε, συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σβετλάνα από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θεωρεί ότι ο ενεργός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αποτελούν κλειδί για να υπάρχει αγαστή συνεργασία. Και έτσι επιτυχάνεται και η λαϊκή συνένεση. Η θέση της βουλγαρικής κυβέρνησης για το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι λοιπόν συνεισφέρουν στην εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων με συνεννόηση. Στη Βουλγαρία οι μισθοί αποφασίζονται ε, με νόμο και ε, ορίζονται από την νομοθεσία. Σύμφωνα με την συνήθη πρακτική, ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής και το βιωτικό επίπεδο στη Βουλγαρία αποφασίζεται από ένα Συμβούλιο Συνεργασίας. Γίνονται σεβαστές οι αρχές της αγοράς και όλες οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα πρότυπα που διέπουν αυτά τα θέματα. Οι μισθοί είναι αντικείμενο συνεννόησης, συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων στη συνέχεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε την ευημερία του πληθυσμού. Αυτό τι σημαίνει. Ότι πάντα προσφεύγουμε στη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό για να είναι η οικονομία μας ανταγωνιστική οι πολιτικές απασχόλησης και οι μισολογικές μετεξελίσσονται, δεν είναι κάτι το στατικό, είναι δυναμική αυτή η διαδικασία και προσπαθούμε να είμαστε και ευέλικτοι. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, δεν επιτρέπονται διακρίσεις βάσει ε, θρησκείας ή οι φύλου. Θα πρέπει όλοι να λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, την ίδια αμοιβή για ίση εργασία. Και αυτή η αρχή πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους τους εργοδότες στη Βουλγαρία. Η κοινωνία μας είναι πάρα πολύ ανεκτική και δεν έχουμε διαφορές μισθολογικές στη Βουλγαρία με βάση αυτά τα κριτήρια. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Τόμας Μαν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει πολύ ένα σημαντικό ε, βήμα από τον Ιούνκερ. Ε, ε, επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο και ο πολίτης μπαίνει στο επίκεντρο. Έγιναν πολλές προσπάθειες, αλλά δυστυχώς όμως σε πολλούς τομείς δεν πέτυχαν. Βλέπουμε ε, ριζοσπαστικοποίηση, βλέπουμε ο κόσμος ε, να ε, πηγαίνει στην άκρα δεξιά. Τι έγινε λοιπόν το σχέδιο Juncker φαίνεται να φροντίζει για επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίστηκε για να εφαρμοστεί η εγγύηση για τους νέους που σε πολλά ε, κράτη δεν ε, εφαρμόστηκε για να δείξουμε στους νέους ότι δεν τους αφήνουμε μόνους τους, αλλά δεν νιώθει κανείς ότι όλα αυτά αποτελούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και κυρία Μανιέ, μια ερώτηση προς εσάς. είχα ε, την δυνατότητα να παρευρεθώ στην ε, Νομισματική Επιτροπή ε, στην Αθήνα και συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Οικονομικών και με άλλους. Το πρόβλημά μας είναι ότι φαίνεται ότι όταν έχουμε μέτρα εξοικονόμησης όλος ο κόσμος λέει ότι αυτό είναι λιτότητα. Όταν όμως έχουμε μέτρα λιτότητας για να υπάρξουν μεταρρυθμιστικά μέτρα και έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα στην Γερμανία. Έχει νιώσει ο κόσμος πόσο ε, σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή να μην περιοριζόμαστε μόνο στην οικονομική πλευρά. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα. Δεν είναι απαραίτητο στη χώρα σας και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει η δυνατότητα μεταρρύθμισης ε, του συστήματος ε, συντάξεών σας. Δεν το κάνουμε αυτό για να παρενοχλήσουμε την Ελλάδα. Πρέπει ο κόσμος να νιώσει πόσο σημαντικό είναι να έχει συντάξεις οι οποίες ε, όμως ε, να είναι βιώσιμες. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδες για το μέλλον στον κόσμο και έχουμε όλες τις καλές προθέσεις, πιστέψτε με. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασιάκος παρακαλώ, από τη Βουλή των Ελλήνων. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε, κύριοι συνάδελφοι. Σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο πρόεδρος ο κ. Μανιός, ήθελα και εγώ να επικεντρώσω τον ενδιαφέρον σας και σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στα πλαίσια της τεράστιας οικονομικής κρίσης της. Το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι σύνθετο και πλήττει ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Τα δεδομένα αυτά επιδεινώνονται σε περίοδο οικονομικής ύφεση μια αναμφισβήτητη και θλιβερή πραγματικότητα για την πατρίδα μου. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργου, δηλαδή ποσοστό 26% ανεργίας. Κυρίως στη χώρα μου έχει επιδεινωθεί ο δείκτης ενεργείας στους νέους που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ε, οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, σταθερότητα και συνοχή. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία μάλιστα εμφανίζουν την Ελλάδα ως τη χώρα με την μεγαλύτερη ανεργία των νέων παγκοσμίω, αγγίζοντας το 51,8%. Και όλα αυτά επιδεινώνονται λόγω της μεγάλης γενικότερης οικονομικής κρίσης μας, καθώς και της εντυνόμενης προσφυγικής κρίσης που πλήττει κυρίω την Ελλάδα λόγω των συνόρων τη, που αποτελούν άλλωστε και σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει έντονη κοινωνική κρίση και η γενικότερη απεσιοδοξία και απόγνωση ε, όπως εκφράζεται από μεγάλο μέρος τη ελληνικής κοινωνίας και κυρίως από τις ευάλωτε κοινωνικές ομάδε. Όλα αυτά τα φαινόμενα οδηγούν σε δοκιμασία και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικέ πρωτοβουλίε μα για την ανακούφιση τη ανεργία των νέων στοχεύουν σε μια βιώσιμη αγορά εργασία για του ε, νέου μέσω τη ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων επιδότηση τη εργασία και όχι τη ανεργία, κατάρτιση και παροχή καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών στη νέα γενιά για την εξέλιξη τη σταδιοδρομία του και την ανέβρεση θέσεων απασχόληση. Η Ελλάδα με αξιοποίηση των πόρων τη ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει σχετικές δράσει που προωθούν την ποιοτική προσφορά της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης, τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα των άνεργων ε, νέων. Παράλληλα, είναι αναγκαία η υιοθέτηση πολιτικών που ενθαρρύνουν τους εργοδότες και υποστηρίζουν τι επιχειρήσει για έγκαιρη διάγνωση των αναγκών του σε σχέση με τι δεξιότητε του ανθρώπινου δυναμικού, για επιμόρφωση των εργαζομένων του, για την παροχή στοχευμένων κινήτρων ικανών να αντισταθμίσουν τα εμπόδια, καθώ και για την ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων. Παρά τι προσπάθειε, δεν έχουν ε, αποδώσει όμω ε, όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε ε, του αναμενόμενου καρπού. Χρειάζεται πράγματι να γίνουν περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει αποτελεσματικότερα τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, γεγονό που αναφυσβήτητα επηρεάζει και τη νέα γενιά. Δεν νοείται, και κλείνω, συλλεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινωνική συνοχή, αλλά χωρί αλληλεγγύη, με τέτοια εντυνόμενη κοινωνική κρίση σε χώρε όπω η Ελλάδα, που κάποια στιγμή κάποτε ήταν στι 10 πρώτε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να θυμάστε το δίλεπτο. Βάντα Κιμαρές από την Πορτογαλία τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα στοιχεία από τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, δείχνουν ε, ότι η λιτότητα στην Ευρώπη δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ότι απλά έχουν πλουτίσει πιο πολύ πλούσιες χώρες. Κάποιοι δείκτες δείχνουν ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά το βιωτικό επίπεδο των Πορτογάλων καθώς και οι συνθήκες εργασίες. Επίσης, έχει αυξηθεί το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες κατά 3%. Η ανεργία έχει φτάσει το 18%, η μακροπρόθεσμη ε, ανεργία έχει πλήξει 4,5 εκατομμύρια ανθρώπων και ε, ο κόσμος απειλείται από την ε, φτώχεια. Πάνω από 400.000 παιδιά και νέοι απειλούνται από αυτήν. Οι καλές θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για το 2016, διότι οι επισφαλές θέσεις εργασίας ε, διονύζουν τις ανισότητες. Οι νέοι εγκαταλείπουν ε, τις πατρίδες τους και μάλιστα οι νέοι που έχουν καλή μόρφωση και εκπαίδευση και αυτό επηρεάζει και τις χώρες γενικά και τις ασφαλίσεις και ε, τις ε, συντάξεις. Δεν είναι δυνατόν ε, να γίνουν μεταρρυθμίσεις χωρίς να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Υπάρχουν πολλοί που ε, ανακατεύονται στο θέμα. Θα πρέπει να σεβαστούμε την αυτονομία των κοινωνικών των κοινωνικών εταίρων και θα πρέπει να υπάρχει τριμερές ε, σύστημα ε, στις χώρες όπου δεν υπάρχει, ώστε να υπάρχει κοινωνική δύναμη. Και στην Πορτογαλία θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές. Επίσης, η ποιότητα της απασχόλησης ε, προκαλεί σημαντικές ε, ανησυχίες, διότι οδηγεί στις ανισότητες ε, και στην φτώχεια. Πρόκειται για μια κατάσταση επικίνδυνη. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για τριπλό α, μάλλον για μονό α στον κοινωνικό τομέα. Η Λάουρα Ατζέα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι αν η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται, είναι αυτή που εμφανίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα Juncker, αν αυτό είναι το πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης, τότε ελπίζω να το ξεπεράσουμε αυτό πολύ γρήγορα, διότι Πραγματικά η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απάνθρωπη θα έλεγα και πάρα πολύ μακριά βρίσκεται από τις πραγματικές κοινωνικές κρίσεις έκτακτης ανάγκης που διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Το παράδειγμα της Ελλάδας είναι εμβληματικό θεωρώ και είναι ξεκάθαρο πώς τελικά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιβλήθηκαν μέσω των προγραμμάτων λιτότητας ισοπαίδωσαν πραγματικά ένα κοινωνικό σύστημα στη χώρα αυτή και είχαν ε, τραγικές συνέπειες για τους πολίτες χωρίς να δημιουργήσουν τα θετικά αποτελέσματα που τίθεται ότι θα δημιουργούσαν και ανταυτού δημιούργησαν μια κοινωνική κρίση. Επομένως, ε, ας μην μιλάμε λοιπόν για αυτό το τριπλό, τετραπλό, πενταπλό α, ας δώσουμε ουσιαστικές, πραγματικές απαντήσεις ε, και ας μην ξεχνάμε τι έκανε τελικά ο πρόεδρος Γιούγκερ και πώς μίλησε για την Ελλάδα. Νομίζω ότι μόνο μέσω κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης μπορούμε να βοηθήσουμε χώρες όπως η Ελλάδα. Έχουμε κρίσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ένα ανθρώπινο πρόσωπο, με μια ανθρώπινη διάσταση. Όλα τα υπόλοιπα είναι και να λόγια τα οποία δεν βοηθούν καθόλου χώρε οι οποίε πραγματικά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα όρια του, στα όρια τη ένδυα και τη πείνα. Ο Φιλιπ Κοντερή, γραμματέα τη Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από τη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η ΟΝΕ δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο ένα σκέλος που είναι το νομισματικό. Η Ευρωζώνη το 2015 ε, διήλθε κάποια ε, κρίση που δεν θα είναι η τελευταία. Αν συνεχίσουν οι ανισορροπίες και οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές και οι κοινωνικές και οι μισθολογικές κυρίως. Εμείς πιστεύουμε ότι η σύγκληση σε αυτούς τους τομείς είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα και μάλιστα σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Το πρόβλημα ποιο είναι ότι το νόμισμα στην Ευρωζώνη δεν είναι πλέον μέσο ανταγωνιστικότητας γιατί δεν μπορείς να κάνεις ανταγωνιστική υποτίμηση. Και η υποτίμηση γίνεται με τους μισθούς εσωτερική. Αυτό είναι ο κίνδυνο. Όταν θέλουν χώρε να είναι ανταγωνιστικέ, επειδή δεν μπορούν να υποτιμούν το νόμισμά του, υποτιμούν του μισθού. Εκεί χρειάζεται πραγματική σύγκληση στι μισθολογικέ πολιτικέ. Βέβαια, οι κοινωνικοί δείκτες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ε, ένα πρώτο στάδιο και βήμα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα και το θέμα του κατώτατου μισθού να είναι στα κοινωνικά δικαιώματα που θα είναι και θα τα προτείνει ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ερχόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε κάθε χώρα να έχει ένα κατώτατο μισθό. Επίσης, στα πλαίσια των συστάσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συστάσεις για την αγορά εργασίας, ειδού να κάνει και άλλες προτάσεις για τα μισθολογικά ζητήματα. Ότι όταν έχει πολύ χαμηλούς μισούς και τέτοια μισθολογική πολιτική, ε, θα πρέπει αυτή να στιγματίζεται για να μην έχουμε dumping μισθολογικό. Και η ανταγωνιστικότητα δεν θα πρέπει να προέρχεται από τους μισθούς. Και τέλος, το να έχουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο μισθών όπου θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και θα έχουν παρουσία μαζί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μας φαίνεται αρκετά ελκυστική, τουλάχιστον πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση για να αντιληφθούμε περισσότερο τι σημασία έχουν οι μισθοί στη γενικότερη μακροοικονομική πολιτική της Ένωσης. Ευχαριστώ. Δύο έχω ακόμα. δεν θα δεχτώ άλλους γιατί έχουμε αρχίσει και πιεζόμαστε από χρόνο για να μπορέσουμε κάπως να προλάβουμε και να παραμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα. Ρίτα Μίλλερ από τη Φιλανδία, παρακαλώ. για δύο λεπτά. Με μικρόφωνο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν αναφερόμαστε στην κοινωνική διάσταση, τότε θα πρέπει να αναφερόμαστε και σε μία ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική αυτή διάσταση και την οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών που ακολουθούμε, πράγμα το οποίο το έχουμε ξεχάσει σε πάρα πολλές χώρες. Βλέπουμε ότι η ανεργία πλήττει πάρα πολλούς πολίτες και ιδίως τους νέους σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθούμε ως κοινωνίες και η ενεργία αυτή οδηγεί τελικά στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλές απειλές. Το προσφυγικό ζήτημα, τους πολλούς ετούντες άσυλο, Επίσης στην αγορά εργασίας βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν τώρα εργασία, οι οποίοι πρέπει με τον έναν τον άλλο τρόπο να ενταχθούν και αναφέρομαι εδώ πέρα πάλι και στους ετούντες άσυλο και γενικότερα στους πρόσφυγες, δεν νομίζω πάντως ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η φυστάμενη αυτή κατάσταση για να οδηγηθούμε τελικά σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων ή σε μια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων δηλαδή. Μια ξεχωριστή αγορά εργασίας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες δηλαδή, οι οποίοι προφανώς θα πληρώνονται με χαμηλότερες αποδοχές. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιγόντως λοιπόν πρέπει να επέμβει από αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονται λοιπόν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερα αποδυναμωμένες στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο σε ένα μοντέλο που θα υφίσταται η δυνατότητα διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους, ανάμεσα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους των εργοδοτών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Έγγελ που είπε ότι τα κοινωνικά θέματα θα πρέπει να ξανατοποθετηθούν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και της αγοράς ε, απασχόλησης. Ε, γι' αυτό θα πρέπει, ε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη, θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να ε, εφαρμόσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος ε, Χέντελ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η νομοθεσία συγκεκριμένων κρατών μελών ε, συμπεριλαμβάνουν κάποιους όρους με πολύ ευρύ ορισμό που επιτρέπουν διάφορες ερμηνείες συχνά υπερβολικές ε, ερμηνείες. Να αναφερθώ σε δύο από τους όρους αυτούς, το κοινωνικό ντάμπινγκ και τις επισφαλείς ε, θέσεις εργασίας. Αυτοί είναι όροι που μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες, ε, συχνά υπερβολικές για να υπάρχει σωστή κατανόηση και για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Καλό θα είναι να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και να αποφεύγουμε όρους που τόσο ασαφείς που να επιτρέπουν τόσες μεγάλες διαφορές στην ερμηνεία. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι εξίσου σαφείς οι όροι που χρησιμοποιούμε και στα 28 κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω υπό το φως των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν να αλλάξουμε τους όρους. Είναι σημαντικό να αυξήσουμε την απασχόληση. Ε, συχνά όμως μιλάμε για καταπολέμηση της ανεργίας όταν μιλάμε για αύξηση της απασχόλησης. Αυτό όμως σημαίνει πώς θα στηρίξουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Η καταπολέμηση της ανεργίας όμως ε, μπορεί να γίνει αντιστρέφοντας το θέμα, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Έτσι είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Έτσι σκεφτόμαστε δηλαδή πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις διάφορες επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ε, προσλάβουν περισσότερους ε, ανθρώπους. Μιλάμε για την διαβίου μάθηση. Οι 20χρονοι τελειώνουν το σχολείο και θέλουν να γίνουν ανεξάρτητοι. Εμείς τους λέμε ότι όχι, χρειάζεστε διαβίου μάθηση. Ας μιλάμε καλύτερα για επαγγελματική εξέλιξη, διότι εάν δώσουμε διαφορετικό όνομα μπορεί αυτό να σημάνει μεγάλη αλλαγή. Ε, συγγνώμη που υπερεύει το χρόνο μου. Ούντο από τη Σλοβενία παρακαλώ. Από την Εθνική Συνέλευση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ε, σε θέση να ε, αντιμετωπίσει την οικονομική ύφεση ε, δεν ήταν έτοιμη να την υποστεί στο βαθμό που την υπέστη. Γιατί τα λέω αυτά. Διότι έχουν επιδεινωθεί οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν για όλες τις τάξεις και τα στρώματα της κοινωνίας. Για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ολοκλήρωση λαών που έχουν τα ίδια δικαιώματα με μια αίσθηση για κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνικά δικαιώματα για όλους. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικά θεμέλια, αλλιώς δεν νοείται ε, πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαλυθεί αν δεν έχει κοινωνικό υπόβαθρο. Το τριπλό κοινωνικό α είναι μια καλή πρόθεση, μια καλή αφετηρία για την πολιτική. Από εκεί και πέρα εγώ χρειάζομαι και επιθυμώ περισσότερες φιλοδοξίες στην υλοποίηση. Για να υπάρχει οικονομία ε, επιτυχής και κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να γίνονται σεβαστά πάντα και παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μου αρέσει αυτή η νομεγκλατούρα, αυτή η ονοματολογία ε, όπου κυριαρχούν ε, τεχνοκράτες με όρους πάρα πολύ σκληρούς, με μέτρα, με στενόμυαλη προσέγγιση και κοντόφθαλμη και μειοπική. Όλα αυτά επιδεινώνουν τη ζωή μας και ε, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Η κοινωνική πολιτική είναι και πολιτική ε, απασχόλησης και οικογενειακή πολιτική και πολιτική για την νεολαία και η πολιτική δεν θα πρέπει συνέχεια να θεωρεί ότι είναι κόστος ε, οι εργαζόμενοι. Μια δαπάνη δηλαδή. Η Γκάμπη Τσίμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα δίλημα. Από τη μια εμείς εδώ ζητούμε όλοι ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη και από την άλλη γνωρίζουμε ακριβώς και πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην κοινωνική πολιτική που είναι κυρίως εθνική πολιτική και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί σήμερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν τίθεται καν το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των αρχών. Δεν το συζητάει καν η Ευρώπη. Γι' αυτό τώρα στις διαπραγματεύσεις, είτε είναι οι συστάσεις αναχώρα, οι εκθέσεις αναχώρα, οι απαιτήσει απέναντι σε κάποιες χώρες που είναι εγώμενες χώρες σε προγράμματα, σε μνημόνια δηλαδή, ε, γίνονται κάποιες ε, μνήες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι σε ευθεία σύγκρουση και απέναντι στα κοινωνικά δικαιώματα. Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς εμείς φανταζόμαστε τα κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική Ευρώπη και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωκοινοβούλιο. Αν εξακολουθούμε να αφήνουμε τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο να ακολουθούν την πολιτική και να μας κάνουν στην άκρη και μην, μην ανακατεύεστε, ε, ασχοληθείτε με τα δικά σας θέματα, είναι θέμα της κυβέρνησης η καταπολέμηση της θα αποτύχουμε γιατί χρειαζόμαστε αλληλεγγύη και αυτή λείπει. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που αξιώνουμε. Δηλαδή όπου και να ζει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να βγει από τη φτώχεια και να ξεφύγει από αυτή. Δεν συζητάμε πια για τους στόχους αυτούς τη στρατηγική τη Λισαβόνας αν θυμάστε. Αυτά έχουν πάει στην άκρη και επιτρέπουμε ε, να ε, παραβιάζονται τα πρότυκα και οι προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Απασχόλησης και Εργασίας, ε, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο κόσμος βυθίζεται στη φτώχεια. Καλό το τριπλό αλφα που ζητάει ο Γιούνκερ, αλλά πότε θα φέρουμε τα κριτήρια, τα συγκεκριμένα και με στόχους μετρήσιμους που μπορούμε όλοι μαζί να ξέρουμε πώς θα φτάσουμε σε αυτούς. Εκεί είναι η κοινή προσπάθεια και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστώ. Αντριάν Σολομών από τη Ρουμανική Βουλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κύριος Μανιός, μετά την οικονομική κρίση σε διάφορες χώρες, τα προγράμματα λιτότητας όχι μόνο δεν έλυσαν τα προβλήματα, αλλά τα κατέστησαν ακόμα πιο σοβαρά. Εμείς, για παράδειγμα, στη Ρουμανία είδαμε ότι ελήφθησαν κάποια πρώτα μέτρα για την κοινωνική οικονομία και το 2010 μειώθηκαν οι αποδοχές κατά 25%. Οι συντάξεις πάγωσαν. Πάγωσε επίσης ο ελάχιστος μισθός, ο κατώτερος μισθός. Τα προβλήματα όμως συνεχίστηκαν και το 2012 μετά υπήρξε μια αύξηση των μισθών και υπήρξε επίσης ε, εκ νέου τιμάριθμος για τις συντάξεις. Αλλά πάλι μετά το 2015 φτάσαμε σε μια οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 4%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν προσαρμόσει κανείς ε, την ε, μισθολογική πολιτική και αν κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, τότε μπορεί να καταλήξει εν τέλει και σε μια κάποια οικονομική ανάπτυξη. Μιλάμε τώρα για αυτά τα συμβούλια ανταγωνιστικότητας, την νέα αυτή ιδέα που ακούσαμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε επίση και την έκθεση των πέντε προέδρων και τη σχετική πρόταση που γίνεται εκεί. Ουσιαστικά όμω πρόκειται εδώ για τον έλεγχο τελικά των μισθών, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο απότερο και βασικό στόχο αυτή τη ιδέα. Κάθε φορά που μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, συμβούλια ανταγωνιστικότητα, ουσιαστικά μιλάμε για ένα μηχανισμό εποπτεία όσον αφορά την εξέλιξη των μισθών που δυστυχώ όμω δεν λαμβάνουν υπόψη τι ιδιάουσε καταστάσει που ισχύουν σε κάθε χώρα και που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι η πρόταση αυτή μπορεί τελικά να επηρεάσει πάλι την όλη διαπραγμάτευση που γίνεται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον καθορισμό των μισθών, τελικά να επηρεάσει την ίδια τη δράση των κοινωνικών εταίρων. Αναφερθήκαμε επίσης και σε διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά είναι επιζήμια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας αν δεν καταφέρουμε να τονώσουμε την εγχώρια ζήτηση. Η εγχώρια όμως ζήτηση θα αυξηθεί μόνο αν μπορεί κανείς να επηρεάσει θετικά όλους τους τομείς της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να προωθηθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την προσφορά και τη ζήτηση και όχι οι πολιτικές αυτές οι οποίες προωθούνται αυτή τη στιγμή που δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο χάσμα σε εθνικό επίπεδο και επίσης πολύ μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι θα πρέπει με έναν τρόπο ευφυή να καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αυξήσουμε την εγχώρια ζήτηση. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο Μοντέρο, από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Αλμπέρτο Μοντέρο. Αλμπέρτο Μοντέρο, από την Ισπανική Βουλή. Ε, Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα κοινωνικό μοντέλο, ευρωπαϊκό εννοώ. Έχουμε κοινή αγορά, έχουμε μια κοινή νομισματική πολιτική και μερικά άλλα κοινά, αλλά όχι κοινό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και δεν μπορεί κανείς να ξεκινάει από μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει αν θέλουμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο που μας ενώνει όλους εδώ. Και μάλιστα να είναι αυτό υπέρ των εργαζομένων ανδρών και γυναικών στις χώρες μας. Ας υποθέσουμε όμως για μια στιγμή ότι υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Τι βλέπουμε και τι βλέπουμε μάλιστα τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα, είναι ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο καταστρέφεται ως συνέπεια των πολιτικών που εφαρμόζονται κατά της κρίσης. Γιατί δημιουργούν διαφορές και μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών προκαλούνται μεγάλες διαφορές διεθνώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εσωτερικό των κρατών, επαναλαμβάνω. Διευρύνονται χάσματα. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικός πυλώνας στην Ευρώπη αν δεν ληφθεί υπόψη τι γίνεται στις αγορές εργασίας. Στη χώρα μου, την Ισπανία, στην αγορά εργασίας τι βλέπουμε. Ένα διπλό σοκ, ένα κραδασμό που ακόμα δεν φαίνεται πώς θα λυθεί. Το ένα είναι ένα ποσοτικό σοκ. Δηλαδή πάνω από 7 χρόνια έχουμε ενεργεία άνω του 20%. Και κάποια στιγμή έχουμε ξεπεράσει και την Ελλάδα, άλλες φορές είμαστε κάτω από την Ελλάδα, χωρίς να έχουμε τη τεράστια ε, κρίση που έπληξε την Ελλάδα και το ΑΕΠ. Πάνω από 45% είναι ενεργία των νέων. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας χωρίς να αυξάνεται το ωράριο εργασίας. Δηλαδή, ε, μοιράζουν την ε, μερική απασχόληση. Και από την άλλη έχουμε και ποιοτική αλλαγή, αυξάνεται η επισφάλεια. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε η σύνταξή τους να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εργαζόμενοι φτωχοί. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την αγορά εργασίας, για τα δικαιώματα, για τη μακροοικονομική ε, προσαρμογή, αλλά να ξέρουμε αυτή η προσαρμογή τι επιπτώσεις έχει στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που ακρηγόρησα. Ο κύριος Φουντούλης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά ακούσαμε ομιλίες ευχολόγια και πάρα πολλά θα. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε εκείνο. Συνηθισμένη λέξη των πολιτικών το θα. Στην πράξη όμως δεν γίνεται τίποτα από αυτά που πραγματικά θα ήταν η διέξοδο στα προβλήματα που πραγματικά μαστίζουν του λαού τη Ευρώπη. Σαν Επιτροπή όλοι μαζί έχουμε διαβουλευτεί, έχουμε συμφωνήσει και έχουμε προτάσει για να βοηθήσουμε να βρεθούν λύσει για θέματα όπω η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία, η ανεργία των νέων. Όμω τι γίνεται στην πράξη. Όλε οι χώρε έχουν τη δυνατότητα ή τη θέληση να εντάξουν στα προγράμματά του αυτέ τι λύσει. Όχι. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από καθεστώ μνημονίων εδώ και πέντε χρόνια. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει ξεχάσει προπολού τι υποσχέσει και τι κόκκινε γραμμέ τη και έχει υποταχθεί πλήρως στι υποχρεώσει έναντι των δανειστών με ένα τρίτο επαχθέστερο μνημόνιο. Σε όλους τους τομείς υπάρχει κατάρρευση. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι στα ύψη, το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας έχει διαλυθεί, όπως και το εθνικό σύστημα υγείας. Η εκμετάλλευση των εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόληση είναι μάστιγα στι μέρε μα. Η αδήλωτη εργασία το ίδιο δεν αρκεί να βάζουμε στόχου εάν δεν υλοποιούνται από τι εθνικέ κυβερνήσει. Η καταστρατήγηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και το, και, κοινωνικό, και το κοινωνικό ντάμπινγκ υπάρχουν. Έχουν καταργηθεί οι συλλογικέ συμβάσει εργασία. Κύριε Μανιέ, δυστυχώ η κυβέρνησή σα δεν δίνει καμία μάχη για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όσα είχατε υποσχεθεί προεκλογικά τα έχετε ξεχάσει και κάνετε ακριβώ τα αντίθετα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες, από τον απλό αγρότη έως τον επιστήμονα, βρίσκονται στον δρόμο. Από θεωρία έχουμε χορτάσει, στην πράξη όμως έχετε αποτύχει. 200.000 νέοι, τα καλύτερα μυαλά της χώρας, επιστήμονες, έχουν φύγει από την Ελλάδα αναζητώντας εργασία σε άλλες χώρες. Πώς θα έχουμε ανάπτυξη με την υπέρμετρη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που τις αναγκάζεται να βάλουν λουκέτο. Μιλήσατε για τις συντάξεις κύριε Μαν στην Ελλάδα Ξεχάσατε να πείτε για την κλοπή των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με το περίφημο PSI που πρότειναν οι δανειστές. Τις 13 μειώσεις στις συντάξεις. Αυτή η λάθος συνταγή της λιτότητας πέντε χρόνια τώρα επιδεινώνει την κατάσταση και δυστυχώς οι θεσμοί και ειδικά η Γερμανία θέλουν να συνεχίσουν την ίδια καταστροφική πολιτική στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Τελευταία ε, Γιάννη Σαντέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός και έχουμε όλη επίγνωση εδώ ότι σε κάποιες χώρες, σε πολλές μάλιστα της Ευρώπης, οι λαοί υποφέρουν από την επισφάλεια, τη φτώχεια και την ανεργία. Θα ήθελα κι εγώ να επιμείνω στην ανάγκη αυτή να είναι πιο κοινωνική η Ευρώπη αυτή η Ευρώπη που υφίσταται τέτοια γενική κατακραυγή σήμερα. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, η ανάγκη να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας ο συνάδελφός μου Έχουμε θεσπίσει κάποια μέτρα και κάποια εργαλεία έχουμε δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και για την ε, ενίσχυση και την ενθάρρυνση της κινητικότητας περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα θέλω να κάνω σήμερα την εξή ερώτηση τελικά. Εντάξει, φέρει κάποια ευθύνη η Ευρώπη, αλλά αυτά τα εργαλεία πώς χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη, πώς αξιοποιούνται τα αξιοποιούν πραγματικά. Οι συστάσεις που γίνονται αναχώρα, συγκεκριμένες, βρίσκουν συνέχεια. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία πραγματικά πρέπει να βρούμε απαντήσεις. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι η ανάγκη να κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πρέπει να φέρουμε αντιμέτωπο τον κοινωνικό πυλώνα με τον οικονομικό. Δεν είναι απέναντι αυτά τα δύο, χρειαζόμαστε και τα δύο. Και ο κοινωνικός πυλώνας θα πρέπει να βασίζεται σε ένα οικονομικό. Και όταν μιλώ για οικονομικό πυλώνα, για μένα σημαίνει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πώς μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να θέλουν να έχουν επιχειρηματικό πνεύμα και να επιχειρούν, να ιδρύουν τις επιχειρήσεις τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι συμπληρωματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό τα κοινωνικά χέρι, χέρι με την επιχείρηση για να μπορούμε να δημιουργούμε πλούτο, θέσεις εργασίας και να ξανάρθουν στην ευρωπαϊκή ιδέα οι πολίτες που την έχουν εγκαταλείψει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτοί ήταν οι συμμετέχοντες και επανέρχομαι στους δύο μιλητές μας. Δυόμιση λεπτά έκαστος παρακαλώ για δευτερολογία. Δυόμιση λεπτά έκαστος για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εθίγησαν πολλά ζητήματα στα οποία βλέπω ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι όχι μόνο η οικονομία αλλά και οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ότι η οικονομική πρόοδος θα πρέπει να συνάδει με την κοινωνική πρόοδο, ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα και συμφωνούμε επίσης ότι ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να διατηρηθεί και ότι θα πρέπει να βελτιωθεί επίσης. Αν δεν εφαρμόζεται σωστά σε κάποια κρατημέλη. Και συμφωνούμε επίσης ότι ε, αν έχουμε μια αγορά δύο ταχυτήτων, τότε σίγουρα είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες αυτές οι οποίες θα ζημιωθούν περισσότερο, τουλάχιστον πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις κοινωνικές πτυχές, τη λεγόμενη κοινωνική διάσταση, ως προς αυτό, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει βασιστεί στο χάρτη του 1989, δηλαδή τον χάρτη των κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ένα χάρτη δηλαδή που εμφανίστηκε πριν από την συνθήκη του Μάστρετ και που στην πράξη όμως δεν υλοποιήθηκε. Εδώ και κάποια χρόνια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία έχει προωθηθεί πολύ περισσότερο η οικονομική πολιτική και η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι αρχικοί θετικοί στόχοι που είχαμε θέσει να μην μπορούν αυτή τη να γιατί υπάρχει μια μείωση της εμπιστοσύνης γενικότερα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε στις πρωτοβουλίες αυτές για τους νέους. Είναι πολύ θετικέ οι πρωτοβουλίε αυτέ, αλλά όντω απαιτείται χρόνο αυτή τη στιγμή, προκειμένου αυτέ να υλοποιηθούν στην πράξη. Νομίζω ότι ε, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μόνο θα μπορούσαμε να δούμε τι ευρωπαϊκέ αυτέ πρωτοβουλίε για του νέου να ελοποιούνται, γιατί επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντε, όπω για παράδειγμα το εκπαιδευτικό σύστημα, τα συστήματα κατάρτιση που υπάρχουν σε κάθε χώρα κτλ. Και βλέπουμε τώρα ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης. Ενδεχομένως να υπάρχει και εκεί μια έλλειψη εμπιστοσύνης και ενδεχομένω να απουσιάζει και το απαραίτητο επίπεδο κοινωνικού διαλόγου. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να επιτρέψουμε στις πρωτοβουλίες αυτές να λειτουργήσουν για ένα κάποιο, χρονικό διάστημα προκειμένου και οι ίδιοι οι πολίτες να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αρχίζει και ενδιαφέρεται περισσότερο για τα κοινωνικά αυτά ζητήματα. Και νομίζω ότι εν τέλει τελικά, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, θα έχουμε σίγουρα κάποιες θετικές επιπτώσεις. η κυρία Ζωζοβιέσκα αναφέρθηκε σε κάτι και όντως παραδέχομαι και εγώ ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέτρα τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία των εκάστοτε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να ελοποιηθούν και να μεταφερθούν τα μέτρα αυτά με τον κατάλληλο τρόπο και να σταλεί τελικά ένα θετικό μήνυμα. Προφανώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα όσον αφορά το ζήτημα αυτό τη μεταφορά και τη υλοποίηση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούν πλέον να έχουν μια πιο κοινωνική Ευρώπη και όχι μόνο μια οικονομική Ευρώπη που είχαμε δει στο παρελθόν. Αυτό από μόνο το αποτελεί ένα πολύ καλό δρόμο, ένα πολύ καλό προσανατολισμό τη κοινοτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαγιό. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ για τη κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο των επιπλέον. Ε, θέλω να ξεκινήσω με μια παρατήρηση ότι θα φύγω από αυτή τη συνεδρίαση εδώ και ενδεχομένως και από την αυριανή περισσότερο αισιόδοξο από, από ό,τι ήμουν μέχρι προχθές. Άκουσα αρκετούς συναδέλφους από διάφορες χώρες διαφορετικών πολιτικών τοποθετήσεων προφανώς οι οποίες έθεσαν σοβαρά ζητήματα υπόψη. Επίσης εκείνο που μου έκανε θετική εντύπωση είναι ότι πολλοί κατάλαβαν πλέον σε διάφορες χώρες ότι το πείραμα της Ελλάδας όχι απλώς απέτυχε, πρέπει να, καθιερωθεί στην ιστορία ως μάθημα προς όλους και μάθημα αποφυγής. Αυτό συνδέεται και με την ερώτηση του συναδέλφου κυρίου Μαν που έχει αυτό το ιστορικό όνομα μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό μας γίνεται μια κριτική γιατί την κάνουμε ο συνάδελφος κ. Φουντούλης είπε ότι είναι ένα από τα πολλά ψέματα που λέμε και είναι όλη η κοινωνία εναντίον μας κάνουμε μεταρρύθμιση ως κυβέρνηση πρώτον στο επίπεδο του θεσμού διότι το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα οφείλουμε να το παραδεχτούμε όχι τώρα στην κρίση, από το 90 γίνονται κουβέντες, ότι ήταν ένα σύστημα τουλάχιστον ανορθόδοξο. Με πολλούς φορείς ασφαλιστικούς όπου ο καθένας ανάλογα την πολιτική του δύναμη και την σύνδεση που είχε με την εκάστοτε κυβέρνηση και εξουσία έπαινε ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ένα σύστημα που μπορούσε ανα πάσα στιγμή μια επιχείρηση τεράστια όπως ήταν η Ολυμπιακή Αεροπορία, όπως ήταν οι τράπεζες να πουλιώνται κλπ. και να διώχνει προώρα τους υπαλλήλους πληρώνοντας πολλά λεφτά για αυτά. Αυτά πρέπει να πληρωθούν κάποτε από τους εργαζόμενους δυστυχώς. Μεταρρύθμιση λέμε λοιπόν εμείς. Ποια ήταν η συμφωνία του καλοκαιριού η οποία μας κάνουν μεγάλη κριτική που την ψηφίσαμε να γλιτώσουμε ένα, οκτα... ένα δις 800 εκατομμύρια ευρώ να μην πάνε από τον προϋπολογισμό στο ασφαλιστικό. Το ένα ήδη το έχει βρει η κυβέρνησή μας με την εδώ και τώρα κατάργηση των πρόωρων συντάξεων. Νομίζει κανείς ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό μέτρο το οποίο το πήραμε χωρίς κόστος. Όλοι που ήξεραν ότι θα ένα 52 χρονών και τους είπαν τα πάνε 65 ή 67 δεν μας θέλουν. Και επίσης έμεινε ένα μικρό ποσό 700 εκατομμύρια. Και είπαμε, έχουμε δύο επιλογές. Να κόψουμε τις συντάξεις για 13η, 14η φορά δεν ξέρω ποια είναι ή να κάνουμε ένα άλλο σύστημα πληρωμών. Και επιλέξαμε το δεύτερο. Οι κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται δεν έχουν άδικο. Γιατί τι έχουν εισπράξει. Έχουν εισπράξει έξι χρόνια μνημονίων. Και αυτά είναι καταστροφικά. Αλλά για να δούμε, είναι μεταρρύθμιση η πρόταση που άκουσα από πολύ επίσημα χείλη και από το Δούνο του και από άλλους να μειώσουμε ξανά τις συντάξεις. Δηλαδή θα μειώσουμε τις συντάξεις, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, γιατρός είμαι. Θα πάρουμε λεφτά από τους συνταξιούχους που παίρνουν λίγα στην Ελλάδα, παίρνουν πολύ κάτω από το μέσο όρο που παίρνουν οι συνταξιούχοι της Ευρωζώνης, θα του τα πάρουμε αυτά τα λίγα λεφτά και θα τα δώσουμε πού, στο δάνειο, στο χρέος, δεν ξέρω πού Αυτά τα λεφτά από πού θα φύγουν? Από την οικονομία. Όταν θα φύγουν τα λεφτά από την οικονομία τι θα γίνει? Θα έχουμε κι άλλη απώλεια θέσεων εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Θα πληγεί και άλλο το ασφαλιστικό. Επομένως μπορεί να λέμε τη λέξη μεταρρύθμιση. Ξέρετε τη ωραία που ακούγεται. Και είναι και ελληνική λέξη. Αλλά αν αυτή είναι σφαγιαστική, ισοπεδωτική, και να πω αυτό και να τελειώσω γιατί μπορεί να έχουν περάσει και τα τρία λεπτά. Ήρθε η κρίση. Κρίση χρέους. Πείτε το όπως θέλετε. Ποιος την πλήρωσε την κρίση στην Ελλάδα. Είμαστε Ευρώπη η οποία νοιάζεται να έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο ή όχι. Αν είμαστε το πρώτο, εμείς προς αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε, πρέπει να δούμε ότι την κρίση την πλήρωσε το 90% τουλάχιστον του ελληνικού λαού και ένα 10% ή δεν πλήρωσε τίποτα ή επωφελήθηκε την κρίση. Μεταρρύθμιση λοιπόν ποια είναι. Να βρούμε τον τρόπο να βάλουμε αυτό το 10% που δεν πλήρωσε τίποτα στην κρίση να το πληρώσει. Αν θέλουμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά θα κυριαρχήσουν απόψεις, δύο ειδών απόψεις. Οι νεοφιλελεύθερες, οι τελείως που καταστρέφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγούν την άκρα δεξιά, συγγνώμη που δείχνω από εδώ, οδηγούν την άκρα δεξιά να παίρνουν πλειοψηφίε και απόψει αριστερέ μεν, αλλά απορριπτικέ τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αριστερέ μεν, γιατί είναι με αριστερή ιδεολογία, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι επιστροφή στα εθνικά κράτη, τα οποία είναι η βάση της όξης των ανταγωνισμών και δύο παγκόσμιων πολέμων που τους γέννησε η Ευρώπη. Να μην γεννήσει και τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο η Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος και η προσπάθεια. Όλοι βλέπουμε τη μεροληπτική, τη μεροληπτική πολιτική των μεγάλων, όχι εθνικών δυνάμεων, των μεγάλων δυνάμεων του κεφαλαίου. Εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε σαφείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και τον Ζωζ και τον Νίκο Τομανιό, για τις αποθετήσεις και τις δηλώσεις και σας όλους για τη συζήτηση. Και όσο αποχωρούν συντεταγμένα οι δύο προηγούμενοι για να έρθουν τα νέα μέλη του πάνελ, θα προσπαθήσω εγώ να κάνω τη μικρή γέφυρα ξέρω ότι πρέπει να είμαστε ακριβείς γιατί μου τα λέει και αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεν θα πρέπει να είμαι επιπόλαιος ε, στην τοποθέτησή μου, αλλά υπάρχει ένα σαφές αριθμητικό στοιχείο. Είναι πάνω από 25, 125 εκατομμύρια σήμερα οι άνθρωποι στην Ευρώπη που βρίσκονται κοντά ή κάτω από το κατόφλι της στόχιας. Και αυτό δεν είναι τυχαίο και είναι και στη στοιχεία του ΩΣΑ. Και στη συζήτησή μας καμιά φορά, πώς να το πω, κοιτάμε μόνο προς μία κατεύθυνση. Η φτώχεια όμως δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζουν οι λεγόμενες χώρες της κρίσης στο Λονδίνο και μόνο το 27% του πληθυσμού ζει κάτω ε, από το κατόφλι της στόχης ή κοντά σε αυτό. Και πάλι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι μαζικό το φαινόμενο η φτώχεια στην Ευρώπη λοιπόν. Και τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι η απόπειρα να φτιάξει την οικονομία εις βάρος των ανθρώπων δεν δουλεύει και πού οδηγεί χάνει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του και δεν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, του προκαλεί ε, αποτροπιασμό, αλλά η πολιτική και καμιά φορά και η ίδια η δημοκρατία και της γυρνάει την πλάτη. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την πολιτική απασχόληση και την κοινωνική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι ως ένα υποπροϊόν ή παραπροϊόν παρακατιανό, όταν έχουμε μια καλύτερη οικονομία ή καλύτερη ανταγωνιστικότητα θα έχεις και μια απώλεια τα κοινωνικά καθόλου. Είναι ένας πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό καλά θα κάναμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε εντατικά και σκληρά και το εθνικό με το ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεχίσει αυτή τη συζήτηση για τις ελάχιστες προδιαγραφές, τις κοινωνικές που να μην είναι, δεν επιτρέπεται να είναι minimum προδιαγραφές ελάχιστες, αλλά κάποιες προδιαγραφές που να δείχνουν το δρόμο προς τα πάνω. Και θα έλεγα ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι η οικονομία δεν μπορεί να βελτιωθεί μόνο με τα κοινωνικά ή μόνο εις βάρος των κοινωνικών. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα και αυτά είναι επενδύσεις και μάλιστα δημόσιες αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Και προσθέτω δουλειές που να μπορεί κανείς να ζει ε, και ιστοδιειναικές και να μην χρειάζεται επιδόματα προνοιακά ή άλλα κρατικά για να ζει. Λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή κατανοώ την πρόταση του Ζαν κλωτ με το ε, σχέδιο επενδύσεων του για την Ευρώπη. Χρειάζεται κοινέ προσπάθειες στην Ευρώπη. Έγινε κάποια κριτική το πρωί, αλλά χρειάζονται συνεργασίες, στρατηγικές υποδομές, έρευνα, ανάπτυξη, ε, καινοτομία. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και σωστά. Για να γίνουν όμως χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε τώρα στο επόμενο πάνελ και καλώς ορίζω θερμότατε την Brigitte van πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ε, των κάτω χωρών. Ε, καλώς ορίσατε θερμά, ευχαριστώ. Και τον κύριο Γιάρο ε, Σαββαντήλ, πρόεδρο επίσης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Τσεχικής Δημοκρατίας. Καλωσορίσατε θερμά στην Επιτροπή μας. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση Ladies First. Παρακαλώ πρώτα η να μας ε, κάνει την πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων Εθνικών Κοινοβουλίων. Το θέμα μας σήμερα είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Θα ήθελα... Για το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στον κόσμο γύρω μας που αλλάζει και τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο των ε, εφιών πόλεων και τον ρόλο των νεοφιών επιχειρήσεων καθώς και το, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ρομποτικής. Όσον αφορά λοιπόν τον κόσμο που αλλάζει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαθίσταται σιγά σιγά. τώρα πια αντί να μιλάμε για αντιμετώπιση της κρίσης μιλάμε για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό το τόνισε και η συζήτηση που είχαμε σήμερα. Αλλά θα πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε ότι η κοινωνία και η αγορά εργασίας δεν είναι ίδια με πριν την κρίση. Έχει αλλάξει αρκετά. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε δουλειά σε περισσότερους ε, άνδρες και γυναίκες. Άλλωστε, αποτελεί έναν από τους στόχους ε, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Χρειάζεται να υπάρξει βελτιωμένη ισορροπία στην αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η ζήτηση να ανταποκρίνεται στην προσφορά και η αντιστοίχηση να γίνεται καλύτερα στις ε, κάτω χώρες, ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες και εργαζόμενοι ε, ενθαρρύνονται να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προετοιμάζουν σωστά τους σπουδαστές για την αγορά εργασίας του μέλλοντος οι σπουδαστές που από νωρίς ε, έχουν αποκτήσει ε, δεξιότητες ε, στις επιχειρήσεις είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το μέλλον και επίσης ενθαρρύνεται η καινοτομία και οι νεοφύση επιχειρήσεις. Για να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους νέους στις αγορές εργασίας, η κυβέρνηση των κάτω χωρών συμφώνησε με οργανώσεις ε, ε, εργοδοτών και εργαζομένων να δημιουργηθούν 10.000 ε, θέσει απασχόληση για τους νέους. Και επίση, πιστεύουμε ότι ένας, ε, μια ιδιαίτερη ρύθμιση μισθολογική για τους νέους ε, ε, ενθαρρύνει την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, η συνεργασία κατά τη γνώμη μας αποτελεί κλειδί για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι κάτω χώρες είναι μικρή χώρα, Έχουμε κάποιες ε, πόλεις, ε, έχουμε... Πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε ε, να έχουμε ανάπτυξη, καινοτομία και απασχόληση και στις περιοχές γύρω από τα αστικά κέντρα. Και το κλειδί βρίσκεται στον σωστό συνδυασμό εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων. Για παράδειγμα, οι Δήμοι να δίνουν άδειε, ε, να βοηθούν στην εξέβρεση του καλύτερου τόπου εγκατάσταση ε, για τι επιχειρήσει, ε, καθώ και τις επενδύσεις στην καινοτομία και την εκπαίδευση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού μας καθώς και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν οι ευφυεί πόλεις, smart cities. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Eindhoven ως καλό παράδειγμα των κάτω χωρών, όπου έχουμε ακριβώς αυτόν τον συνδυασμό. Είναι μια πόλη στα νότια των κάτω χωρών. Ε, έχουμε εκεί σημαντικές ε, μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η Philips. Ε, το 2011 η περιφέρεια γύρω από την πόλη του Eindhoven θεωρήθηκε η πιο ευφυής περιφέρεια στον κόσμο από το σχετικό φόρουμ και νεοφυείς επιχειρήσεις ε, στην περιφέρεια αυτή αλλά και ε, στο υπόλοιπο της χώρας ε, αποτελούν σημαντική κινητήριο δύναμη της καινοτομία. Όπως άλλωστε και οι ευφυείς πόλεις και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει η διακυβέρνηση όλων των επιπέδων να συνεργάζεται στενά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους επιχειρηματίες. Όσον αφορά τη σημασία των νεφιών επιχειρήσεων, όλοι γνωρίζουμε και υπόθηκε και αυτό ότι είναι πολύ σημαντικέ οι οικογενειακέ επιχειρήσει και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, όπω άλλωστε και οι νεοφυεί επιχειρήσει. Ε, μία σχετική πρωτοβουλία είναι η πρωτοβουλία ΔΕΛΤΑ ε, για τι επιχειρήσει αυτέ. Ε, ήταν πρωτοβουλία τη πρώην Επιτρόπου Νέλη Κρούς και στόχο είχε να δημιουργήσει τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε για τι νέε επιχειρήσει Μέσα σε λίγους μήνες οργανώθηκε το Φεστιβάλ Νεοφιών Επιχειρήσεων όπου οι επενδυτές και οι ε, και επιχειρηματίες θα συναντηθούν. Θα συμμετέχει ο CEO της Apple, Tim Cook, της Uber επίσης, ο κύριος και της Alibaba, ο Jack May. Αναμφίβολα θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να εμπνεύσουν και τους δικούς μας επιχειρηματίες. Πριν λίγες εβδομάδες επισκέφθηκε τη χώρα μας ο Bill Gates και είχε συναντήσεις με διάφορες νεοφύσεις επιχειρήσεις αλλά και με μέλη του Ολλανδικού Κοινοβουλίου για την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία και οι νέες επιχειρήσεις να λάβουν εναλλακτική χρηματοδότηση διότι είναι σημαντική η χρηματοδότηση για τις νέες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν μπορούμε να εμπνεύσουμε τους νέους, ε, να ε, τους βοηθήσουμε να δικτυωθούν και να τους βοηθήσουμε να βρουν χρηματοδότηση. Στην ε, Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων ε, πρόσφατα ε, υιοθετήσαμε θεματολόγιο που περιέχει 43 προτάσεις για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη η γνώση ε, και η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ και την έννοια του crowdfunding, που είναι εναλλακτικός ε, και πολλά υποσχόμενος τρόπος ε, χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων και έτσι δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Οργανώθηκε στρογγυλή τράπεζα για το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και οι βουλευτές συζήτησαν τρόπους να βελτιώσουν τις συνθήκες ε, για τις επιχειρήσεις ε, με το crowdfunding. Έτσι το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει το ρόλο του ε, στηρίζοντας νέες και καινοτόμες ιδέες. Και τέλος θέλω να αναφερθώ στην ρομποτική. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να επωφελούμαστε από την καινοτομία θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος ε, ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο. Οι τεχνικές εξελίξεις ε, και η εξέλιξη των ρομπότ ε, θα επηρεάσουν την οικονομία μας και ιδιαίτερα την αγορά εργασίας. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολλανδικής Βουλής Αντιπροσώπων αποφάσισε να δράσει προορατικά, να προορατικά και να αναθέσει έρευνα σχετικά με το τι μπορούμε να περιμένουμε από διάφορες εξελίξεις της τεχνολογίας. Η έρευνα αυτή εξέτασε σημαντικές ε, εξελίξεις ε, στην τεχνολογία του παρελθόντος. Ε, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Έτσι μπορούμε να μαντέψουμε ποιοι θα βγουν κερδισμένοι αυτή τη φορά και ποιοι πιθανότατα να βγουν χαμένοι. Έτσι θα μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσουμε. ερωτήματα όπως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε όσον αφορά ε, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να επιλέξουν τον κατάλληλο κλάδο. Για παράδειγμα, να μην σπουδάζουν όλη ψυχολογία, αλλά και ε, τεχνολογίες ε, της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Επίσης, επαγγελματική κατάρτιση για τους νέους ή νομική προστασία για κάποιες ομάδες εργαζομένων που μπορεί να κινδυνεύουν από τις εξελίξεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που μπορούμε να κάνουμε και η Επιτροπή στην οποία εργάζομαι εγώ στο ε, Ολλανδικό Κοινοβούλιο ασχολείται με τα θέματα αυτά. Τέλος, όπως ανέφερα και πριν, η συνεργασία μεταξύ μας, να εμπνέει το ένας από τον άλλον, ε, να προκαλεί ο ένας τον άλλον, ε, νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα. το να αναλαμβάνει κανείς δράση, το να αναλαμβάνει τις ευθύνες στη χώρα του και ε, να μην φοβάται να λάβει δύσκολες αποφάσεις είναι κλειδιά για την επιτυχία στο μέλλον ώστε να έχουμε ανταγωνιστικές χώρες, ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες. Πιστεύουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει διακοινοβουλευτική συνεργασία με ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, όχι μόνο μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά και ανάμεσα στους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και τους Ευρωβουλευτές. Έτσι μπορούμε όχι μόνο να ενισχύσουμε τον δημοκρατικό έλεγχο, αλλά να υποφεληθούμε ο ένας από τις ε, ιδέες του άλλου και να μάθουμε ένας από τα λάθη του άλλου. Ίσως να μαθαίνει κανείς περισσότερο από τα λάθη. Εγώ ήμουν στο παρελθόν επιχειρηματίας και όταν αποτυγχάνει κανείς μαθαίνει περισσότερα. Ελπίζω να συνέβαλα στο στόχο αυτό και προσβλέπω ε, στις, σε αυτά που μπορώ να μάθω από τους συναδέλφους και θα ήθελα να ακούσω τις παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπριγκίτε Φαντεμπούρχ, για την πρώτη αυτή τοποθέτηση. Μου είπαν ότι ο Γιάρος ε, Ζαβαντήλ δεν είναι απλός πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά επί σειρά ετών ήταν επικεφαλής συνδικαλιστικής οργάνωσης ε, της αντίστοιχης ΓΕΣΕ της Τσεχίας. και πάλι. Και μια που είστε και συνδικαλιστή, εγώ χαίρομαι ακόμα περισσότερο που έχω την ευκαιρία να σας καλωσορίσω. Λοιπόν, Γιάροσλαβ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Τόμας. Κάθομαι δίπλα στον κοινωνικό εχθρό μου, θα έλεγα. Δίπλα σε επιχειρηματία. Έτσι δεν είναι. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Αυτό είχε πει ο Άμλετ πριν από πάρα πολλούς αιώνες. Στην Τσεχία είχαμε συγκεκριμένες εξελίξεις κάτι διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση. Πολλά πράγματα όμως δεν ευωδόθηκαν, πολλά πράγματα δεν οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα και κληθήκαμε να αναρωτηθούμε γιατί. Αν δεν κάνω λάθος, ο Φιλανδός συνάδελφος μας είπε ότι κοινωνία και οικονομία θα πρέπει να συνάδουν, να συμπορεύονται. Εμείς στο παρελθόν είχαμε πει ότι θα πρέπει να έχουμε μία κοινωνική οικονομία, μία ισορροπημένη λύση η οποία θα συνδύαζε τόσο οικονομική πολιτική όσο και μία δίκαιη κοινωνική πολιτική. Το 2009, όταν έφτασε η οικονομική κρίση και στη δική μου τη χώρα, ξεκίνησε μία πολιτική λιτότητος. Σταμάτησαν επενδύσεις, οι μισθοί, οι συντάξεις, γενικότερα οι αποδοχές στη χώρα μου, πάγωσαν ήταν θύμα της πολιτικής λιτότητας και συνειδητοποίησαμε βέβαια ότι δεν θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να διηγηθούμε σε ευημερία. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνησή μας συνέχισε αυτή την πολιτική λιτότητας. Το 2012 λοιπόν, μολονότι ε, χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Σλοβακία ήδη είχαν οδηγηθεί σε μια κάποια οικονομική ανάκαμψη και είχαν ε, ανάπτυξη της τάξης του 1,5 ακόμα και 3% του ΑΕΠ, εμείς στην Τσεχία τη χρονιά εκείνη είχαμε αρνητική ανάπτυξη. Και αυτό εξαιτία της πολύ σκληρής πολιτικής λιτότητας που ακολουθούσε η κυβέρνηση στη χώρα μου. Περίπου 600.000 600 ήταν οι άνεργοι, δηλαδή περίπου το 10% του ενεργού πληθυσμού. Στη συνέχεια, κληθήκαμε βέβαια να λάβουμε κάποιες αποφάσεις που θα θεράπευαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν, ή πιο συγκεκριμένα το 2015, η τσεχική δημοκρατία είχε μια ανάπτυξη της τάξης του 4,4% σε σχέση με το ΑΕΠΑ. Αναφέρουμε πάντα στοιχεία του 2015. Η ενεργεία μειώθηκε κατά 140.000 λιγότερους ανέργους και αυτό γιατί γίνανε πολύ σημαντικές επενδύσεις. Και γιατί επίσης ανέλαβαν ενεργή δράση και τα γραφεία εξέβρασης εργασίας. Είχαμε νέο προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες απασχόλησης και ως αποτέλεσμα είχαν πλέον την ε, δυνατότητα οι υπηρεσίες αυτές, τα γραφεία αυτά, να βοηθήσουν ε, τους ανθρώπους να βρούνε μια θέση απασχόλησης. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η ενεργία έχει μειωθεί στο 6%, ένα ποσοστό το οποίο είναι θετικό, αν δούμε τη γενικότερη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου όπως ακούσαμε σήμερα υπάρχουν χώρες που έχουν ανεργία της τάξης του 20% ή ακόμα υψηλότερα ποσοστά, ιδίως όσον αφορά την ενεργία των νέων. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν απασχόλησης σε βρέσος εργασίας στην Τσεχία υιοθέτησαν πολλά θετικά μέτρα. Για παράδειγμα προσπάθησαν να δώσουν κίνητρα χρηματοδοτικά μέσω επιδοτήσεων σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες οι οποίοι θα αναλάμβαναν να απασχολήσουν νέους αλλά και ηλικιωμένους εργαζομένους, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται πάνω από την ηλικία των 50 ετών. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι η νεανική ανεργία είναι μία από τις χειρότερες μορφές ανεργίας και βλέπουμε τώρα ότι γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλονται προσπάθειες για να καταπολεμηθεί αυτή η νεανική ανεργία. Έχει λοιπόν σημειωθεί μια κάποια πρόοδο, σίγουρα. Αλλά ας δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Εμείς έχουμε, ή μάλλον βλέπουμε ότι έχουμε νεανική ανεργία, έχουμε διαρθρωτική ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα, δεν έχουμε τι απαραίτητε πληροφορίε για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα τη κατάσταση. Όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό το οποίο συνειδητοποιώ είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη σύμπνοια και ένα γενικότερο πνεύμα συνεργασία για τα ζητήματα αυτά. Εμεί από το 2004 και μετά ως ειδικαλιστική οργάνωση είχαμε προφανώς προωθεί την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πιο έντονη συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε βέβαια η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν, αλλά είμαστε ακόμα πεπισμένοι ότι πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη. Στην Τσεχία πιο συγκεκριμένα μας απασχολεί προφανώς και το ζήτημα της μετανάστευσης. Δεν μας έχει πλήξει ιδιαίτερα ακόμα το προσφυγικό ζήτημα. Είμαστε μια χώρα διέλευσης περισσότερο θα έλεγα. Βλέπουμε απλώ μετανάστες οι οποίοι οδεύουν περισσότερο προ τη Γερμανία, προφανώς επειδή θεωρούν ότι εκεί πέρα έχουν καλύτερες ε, ευκαιρίες ε, απασχόλησης από ό,τι στην Τσεχία. Το ερώτημα όμω που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι τι μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διακινδυνεύουν τα πάντα και πολλές φορές κινδυνεύει και η ίδια η ζωή τους. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί τελικά καταλήγουν να είναι τόσο επιλεκτικοί. Για ποιο λόγο δεύουν κυρίως προς τη Γερμανία. Για ποιο λόγο δεν παραμένουν στην Τσεχία που είναι και αυτή μια ασφαλής χώρα. Ενδεχομένω λοιπόν επιλέγουν οι μετανάστε στι χώρε εκείνε που έχουν καλύτερα συστήματα κοινωνική ασφάλιση. Τίθεται πάντω το ερώτημα. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είστε ένα θεσμικό όργανο αρκετά πολύπλοκο και δεν νομίζω ότι πρόκειται να απλοποιηθεί η δομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ έχω κυρίω εμπειρία από το εθνικό μου το κοινοβούλιο, το οποίο είναι πολύ μικρό αλλά εξίσου πολύπλοκο και αυτό στη λειτουργία του και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανεί σε συνένεση. Στο δικό μου το κοινοβούλιο που είναι μικρό, πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο κοινοβούλιο όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά συγχαρητήρια εφόσον καταφέρατε και καταλήγετε τελικά σε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Εμείς θέλαμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει να πράξουμε και στο μέλλον. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές που θα δημιουργούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικές που θα δημιουργούν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον και για τη λειτουργία των ίδιων των εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου αυτά με τη σειρά τους να μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης επιτόπου σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Μιλάμε όλο και περισσότερο για ανταγωνιστικότητα, για συμβούλια ανταγωνιστικότητας. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι όρο τελικά θα επιλέξουμε. Πρέπει ουσιαστικά να εφίσταται ένας τέτοιος θεσμός. Αλλά προσοχή, θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη σύμπνοια, συνεργασία και ένα κλίμα κατανόησης ανάμεσα σε κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους. Αν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο δεν πάμε πουθενά. Νομίζω λοιπόν ότι οι κυβερνήσεις, οι πολιτικά ηθήνοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον διαλόγου μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, οργανώσεων εκπροσώπησης των εργοδοτών. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να υφίσταται. Αν δεν υφίσταται ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον, χάνουμε τα πάντα, θεωρώ. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Ένα πολύ καλό φίλο μου από την Ελλάδα τον έχουμε σήμερα εδώ πέρα στην αίθουσα. Έχουμε κάνει εκτενέστατη συζητήσει για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει όμω να φερόμαστε σε μονομένε μονοχώρε. Τα ζητήματα αυτά αφορούν όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, διαλλακτικοί και θα πρέπει να εστιαζόμαστε στην αλήθεια. Ακόμα και δεν μα βολεύει πολλέ φορέ η αλήθεια ή δεν μα αρέσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στη σωστή διάσταση των πραγμάτων. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολυσχηδή προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να εργαστούμε στα εθνικά μας κοινοβούλια. Είτε είμαι πάντως εθνικός βουλευτής, είτε είμαι ευρωβουλευτής, νομίζω ότι πρέπει ουσιαστικά να έχω πλέον τους ίδιους στόχους. Νομίζω ότι όλοι, είτε από τις χώρες μας, είτε εδώ στις Βρυξέλλες, μπορούμε να συμβάλλουμε προκειμένου να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη. Ένα στόχος ο οποίος τελικά δεν είναι εύκολος. Ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθε είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μεταλλορύχοι, μεταλλουργοί στι στις Βρυξέλλες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν κυρίως για το άνοιγμα που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κίνα. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε ευνοϊκέ συνθήκε εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατάλληλο περιβάλλον ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λειτουργούμε τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπουμε τελικά ότι οι ίδιες συνθήκες εργασίας δεν υφίστανται σε μια χώρα ανατολική όπως η, Κίνα. Ξέρετε επίσης ότι έχουμε ένα διεθνή οργανισμό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, στον οποίο συμμετέχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και στον οποίο από κοινού μπορούμε να προασπίσουμε ορισμένες από τις εργασιακές συνθήκες που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω για παράδειγμα ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα της χαλιβουργίας στη χώρα μου. Βλέπω τι υποδομή, τι εξοπλισμό έχουμε εμεί στην Τσεχία και τι εξοπλισμό έχουν για παράδειγμα στην Ινδία. Μιλάμε για δύο καταστάσει οι οποίε δεν μπορούν να συγκριθούν, είναι εντελώ διαφορετικέ. Το κόστο εργασία, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα και πολύπλοκο μάλιστα ζήτημα. Το θέμα της παιδικής επίσης εργασίας. Εμείς επί της αρχής προφανώς είμαστε κατά της παιδικής εργασίας. Ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ινδία ή το Μπαγκλαντές όπου τα παιδιά εργάζονται ή αναγκάζονται να εργαστούν προκειμένου να συμβάλλουν και αυτά βιοποριστικά στη ζωή των οικογενειών τους. Αν ανοίξουμε όμως τώρα εμείς τα σύνορά μας και να επιτρέψουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αν μη τι άλλο οφείλουμε να επιβάλλουμε τους δικούς μας τους κανόνες, τους εργασιακούς, τη δική μας την επικράτεια. Να ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για όλους αυτούς τους μετανάστες που έχουν έρθει, που προτίθενται να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το απότερο θεωρώ καθήκον μας. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτού οι οποίοι νομίμως έρχονται στις χώρες μας για να ζητήσουν μια θέση απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του εργασιακού δικαίου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, Γιάροσλαβ. Τώρα είπε τόσε λέξεις, τέσσερις έννοιε που μπαίνω στον πειρασμό να κάνω και εγώ τοποθέτηση, πράγμα που δεν θα πράξω, μην ανησυχείτε. Ε, επτά συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και εγώ είμαι κοδεσπότης και πρέπει να συντονίσω. Όχι χέρια, μόνο με ε, το κίτρινο αυτό χαρτάκι, αγαπητοί συνάδελφοι. Μόνο αυτό το κίτρινο, αλλιώς δεν μπαίνει το λόγο κανείς. Έχω πάρα πολύ αυστηρές εντολές. Λοιπόν, όποιος θέλει να ζητήσει το λόγο, παρακαλώ συμπληρώσει αυτό το κίτρινο χαρτί για να το ζητήσει επίσημα και όχι με τα μπελάκια και ονόματα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Από την Πολωνία, το Μίτσοσλαφ Αγουστίν από την Πολωνική Βουλή. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πολλά ακούσαμε και πολλά συναισθηματικά φορτισμένα, διότι η κρίση έχει πολλές κοινωνικές επιπτώσεις και συνήθως εκεί εστιάζουμε και καμιά φορά ξεχνάμε τις τεράστιες αυτές διαδικασίες και διεργασίες που συμβαίνουν ανεξαρτήτως ε, των τρέχουσών εξελίξεων. Δηλαδή ξεχνάμε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη ή το νέο κοινωνικό θεματολόγιο, ε, αλλά υπάρχουν και η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή, η γύρανση του πληθυσμού, η τεχνολογική πρόοδος και θα ήθελα να αναφερθώ στη γύρανση του πληθυσμού παραδόξως ως χώρο επένδυσης. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε στην Ευρώπη να το θεωρούμε μόνο βάρος, ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον προϋπολογισμό. Βεβαίως και κοστίζει, αλλά μπορεί να είναι και επένδυση. Τι σημαίνει αυτό, ότι με τα περιορισμένα μέσα και πόρους που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε τις κοινωνικές αλλαγές. Είναι παράδοξο αυτό. Στην Ευρώπη έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τεράστιο αριθμό ανέργων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ένας καλός τρόπος να το ξεπεράσουμε είναι να αναπτύξουμε τις νέες αγορές που δημιουργούν εργασία. Που δημιουργούν δουλειές. Ε, μία από αυτές τις αγορές ή ένας κλάδος, εν πάση περιπτώσει, που καμιά φορά ξεχνάμε και πολύ συχνά, είναι η ενας κλαδος σε παση περιπτωσει που καμια φορα αυτή των υπηρεσιών φροντίδας προς τους ηλικιωμένους. Ε, ε, είναι ένα καλός χώρος και για καινοτομία και για επενδύσεις. Και εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε εκατομμύρια θέσεων εργασίας για ανθρώπους που φροντίζουν τους άλλους. Με προσόντα, με δεξιότητες ε, για ανθρώπους που δεν είναι πλέον ανεξάρτητοι. Υπάρχουν χώρες που κάνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Κάθε μια χώρα κάνει ό,τι μπορεί και η Πολωνία διότι το βλέπουμε αυτό ως ευκαιρία για να δημιουργήσουμε 400.000 παρακαλώ θέσεις εργασίας. Και τέλος θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Μπριγκίτ Φαντενμπερκ. Εγώ είμαι από την Κίο στην Πολωνία, ε, όπου έχουμε τέσσερα εργοστάσια της Philips. Πάμε συχνά στο Αιτχόβεν και θα δημιουργήσουμε και εμείς μια ευφυή πόλη στη δική μου περιφέρεια. Τέσσερα εργοστάσια Philips έχετε στην Πολωνία. Σέβας. Ε, Ράσου, ο συνάδελφος από τη Λετωνία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι οι μισοί ομιλητέ ε, είναι Έλληνες και οι άλλοι μισοί μιλάνε για την Ελλάδα. Αλλά κρίση είχαμε και στη Λετωνία. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποια ζητήματα που λειτουργούν καλά, κατά τη δική μας γνώμη. Είχαμε μακροσκελή συζήτηση για τις επενδύσεις πριν κάποιο διάστημα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και τη σημασία της ε, συμμετοχικής και βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι σημαντικό οι επενδύσεις να δημιουργούν νέες και υψηλής ποιότητας ε, θέσεις εργασίας ε, για ε, την προώθηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και την καταπολέμηση της φτώχειας. Όπως και ο προλαλής σας είπε από την Πολωνία. Άλλωστε, το ίδιο μπορεί να υποθεί σχετικά με τη βελτίωση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και αυτό μας βοήθησε πολύ να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με την κοινωνική ένταξη και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Στη Λετωνία βλέπουμε άμεση σχέση ανάμεσα στους δείχτες της αγοράς εργασίας και το επίπεδο ε, της μόρφωσης των εργαζομένων. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο, τόσο καλύτερη η θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας και πιστεύω ότι η ε, υψηλή σε ποιότητα θέσει εργασίας που να βασίζονται ακριβώς σε, σε σωστή μόρφωση μπορούν ε, να βελτιώσουν την κατάσταση. Η σημαντική λοιπόν στη συζήτησή μας είναι η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης. Ε, θα πρέπει Επίσης να γίνεται σωστή ε, αντιστοίχηση μεταξύ δεξιοτήτων ε, και θέσεων εργασίας. Πολύ ενδιαφέρον ε, στα δεδομένα από το τρίτο τρίμηνο τρίμηνο του 2014 δείχνει ότι η ανεργία των γυναικών είναι 8,6% ενώ των ανδρών είναι 11%. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δείχνει τουλάχιστον ότι όσον αφορά την ισότητα τα πάμε καλά. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Δεν έχει αλλάξει το καθεστώς. Δύο λεπτά έχει ο καθένας. Αλεξάνδρου Πέτρου Φρετεάν, παρακαλώ. Από την Ρουμανία, παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές για μένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ταυτόχρονες κρίσεις. Σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο έχουμε την αργία, τον πληθωρισμό, ε, το θέμα μετανάστευση, θέματα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αξιοπιστία και ε, αλληλεγγύη για να βελτιώσουμε την ε, εμπιστοσύνη από πλευράς των πολιτών μας ε, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την οικονομία μας ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες. Έτσι ε, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα που υπάρχει διαπιστώνουμε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις και καλύτερη βελτίωση στην ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα αποτελέσει καλή λύση για να βελτιωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να ε, οικοδομηθούν ε, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Και θα πρέπει οι πόροι του προϋπολογισμού να χρησιμοποιηθούν σε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα πρέπει να δώσουμε και κίνητρα στην ε, στις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπιστεύονται περισσότερο τις ε, δημόσιες πολιτικές και, τα, και τους θεσμούς. Χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα και να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ε, κοινό συμφέρον και στο συμφέρον όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Η Λάουρα Ατζέα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενάμιση ε, χρόνο έχει περάσει στη νέα αυτή θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε αναλογιστεί κατά καιρού πραγματικά ποιε πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων απασχόληση αν μπορούμε να έχουμε έναν νέο επαναπροσανατολισμό όσον αφορά τις δεξιότητες, αν μπορούμε να επενδύσουμε σε κάποιους νέους τομείς, όπως για παράδειγμα η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία για παράδειγμα. Όλα αυτά θεωρητικά είναι πολύ ωραία και πολύ δίκαια. Αλλά στην πράξη αυτό που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τώρα είναι ότι ε, βλέπουμε ότι φύστανται πάρα πολλοί κίνδυνοι που έχουν να κάνουν ε, από κάποιες μακρινές μας πραγματικότητες που ζυγώνουν όμως όλο και περισσότερο. Αυτό το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει στην Κίνα το καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην πράξη ουσιαστικά θα εκμηδενήσει οποιαδήποτε δική μας πρόθεση, θεωρία, τοποθέτηση, πρωτοβουλία προκειμένου να αυξήσουμε την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά θα ζημιωθούμε, θα ασκηθεί πάνω μας όλη αυτή η έντονη παραγωγική πίεση της Κίνας και πραγματικά δεν θα ξέρουμε πώς και δεν θα μπορέσουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο παραγωγικός μας ιστός θα διαλυθεί. Νομίζω ότι έχουμε προσπαθήσει στο παρελθόν να προωθήσουμε να επικοδομητικά τη δική μας την παραγωγή, αλλά δεν το καταφέρουμε απέναντι στην Κίνα. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα τεράστιο κοινωνικό ντάμπινγκ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό κοινωνικό ντάμπινγκ όταν η Κίνα μπει στη δική μας την αγορά. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να θέσουμε. Μπορούμε να μιλάμε προφανώς για απασχόληση, για βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τεράστιους κινδύνους σαν αυτόν που θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ούρο από την Σλοβενία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Εδώ τώρα εμείς συζητάμε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι πραγματικά από τα βασικά καθήκοντα οποιασδήποτε πολιτικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να είναι ποτέ ούτε υποπροϊόν ούτε παραπροϊόν όπως είπατε εσείς πρόεδρε. Η παράπλευρη απώλεια. Όλοι μας θέλουμε πλήρη απασχόληση και 0% ανεργία. Αυτό στην πράξη δεν είναι ποτέ δυνατό. Μπορεί στη θεωρία να ακούγεται καλό. Θέλουμε να ε, καταργήσουμε επίσης τις επισφαλείς μορφές εργασίας και ε, τη μερική απασχόληση, την αναγκαστική μερική απασχόληση που δεν ε, παρέχει καμία προοπτική ούτε κοινωνική ασφάλεια. όταν πετυχαίνει η ε, πολιτική της εργασίας χρειάζεται λιγότερη ενέργεια και λιγότερες επενδύσεις η ε, πολιτική της κοινωνικής πρόνοιας για να φτάσουμε στο τριπλό α που μας απασχόλησε προηγουμένως, το κοινωνικό. Βεβαίως, κάθε κράτος και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβληματιστούν για το τι θέσεις εργασίας θέλουμε, τι δουλειές θέλουμε να ανοίγουν στην Ευρώπη. Πάντως ένα είναι γεγονός ότι όλοι που εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας για την ίδια δουλειά θα πρέπει να παίρνουν τον ίδιο μισθό και μάλιστα δίκαιο και σωστό. Ορισμένοι μιλούν για την ειδίκευση. Εντάξει, είναι καλή αυτή και σημαντική, αλλά θα πρέπει να μιλάμε και για την ανάπτυξη των περιφερειών μας. Ε, καλή ειδίκευση και η ευφυής ε, περιφέρειες, αλλά πρέπει να συνδυάζουμε σε αυτό τον τομέα ε, όλους τους ε, κλάδους της οικονομίας. Κάτι άλλο που πρέπει να προωθήσουμε είναι η συνεργασία με τα πανεπιστήμια, διότι θέλουμε να έχουμε καλές ποιοτικέ θέσεις εργασίας που να παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα, από την Κύπρο, ε, η κυρία Σκέβη Κουμά. Yeah. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με την θέση του Προέδρου της Κομισιόν ε, για τις νέες θέσεις εργασίας ε, ότι θα πρέπει να τις δημιουργούν οι επιχειρήσεις και όχι οι κυβερνήσεις ή οι θεσμοί. Αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι μια παλιά θέση η οποία έχει αποδειχτεί στην πορεία ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Και ήθελα να σχολιάσω έτσι και παρατηρήσεις που έγιναν στην προηγούμενη σύνοδο, όπου γινόταν αναφορά παραδείγματο χάρη στη διαβίου μάθηση, που όλοι κατανοούμε ότι πρόκειται για μέτρα συνεχούς μετεκπαίδευση των εργαζομένων για να μπορούν να βρουν κάποια αναπασχόληση. Μιλούμε όλοι για την τοποθέτηση ανέργων σε εταιρείε και ότι οι εταιρείε θα πρέπει να αυξήσουν τι θέσει στι επιχειρήσει του. Όλα αυτά μιλούμε για μερικής απασχόλησης ε, εργασίες, ε, όχι μόνιμες, πλήρους εκμετάλλευσης και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη διάσταση μόνιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Και θα ήθελα εδώ να σχολιάσω τη θέση της αρμόδιας επιτρόπου, η οποία είχε παλιά ε, θέση της και αναφερόταν σε ίσες ευκαιρίες για όλους ενώ τώρα μιλά για αξιοπρεπείς ευκαιρίες για όλους γιατί όλοι έχουν κατανοήσει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες γι' αυτό στοχεύουμε στις αξιοπρεπείς τουλάχιστον. Να πω ότι η προσπάθεια για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεστε ότι στοχεύει στη μείωση των μισθών και από εκεί ξεκινούν όλα. Ε, να κάνω έτσι μόνο μία αναφορά ότι στην Κύπρο το 2015 είχαμε 15.000 εντάλματα φυλάκισης για οφειλές προ τι προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις ε, σε άλλα ε, φόρους, ΦΠΑ και άλλα, τα οποία αναστάληκαν που υποχρεώθηκε το κράτο μέσω του Γενικού Εισαγγελία, να δώσει αναστολή γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Είναι κυρίω μικρομεσαίε επιχειρήσει που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του και οδηγούνταν στη φυλακή οι επιχειρηματίε ή οι εργαζόμενοι ανάλογα. Έτσι δεν μπορούμε να συζητούμε άλλον παρά το ότι θα πρέπει να γίνουν δημόσιες επενδύσεις για να μπορούμε να προσβλέπουμε σε βιώσιμες και ποιοτικέ θέσεις εργασίας που θα, θα στηρίζουν και το κοινωνικό κράτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τάνια Γκονσάλης Πένιας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια υφίσταται μείωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών της και πάρα πολύ σημαντική επιδείνωση και αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε θεομηνία, ούτε γιατί έτσι μας ήρθε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα και καρπός πολιτικών αποφάσεων. Διαχείριση της κρίσης που βασίζεται στην υποτίμηση των δημοσίων υπηρεσιών και στην υποβάθμιση και επιδείνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι καρπός πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν από τούτα εδώ τα θεσμικά όργανα. Είναι δράμα, τραγωδία είναι νεανική ανεργία. Πολύ ακούστηκε σήμερα και πλήττει την Ευρώπη όλο και περισσότερο σε χώρες όπως η Ισπανία. Η Ισπανία είναι πρώτη, πάνω από 50% ενεργεία των νέων, πρωτοστατή. Και μπροστά σε αυτό το δράμα και την τραγωδία, οι λύσεις που δίνουμε ποιες είναι. Είναι μπαλώματα, ε, δεν λύνουν την κατάσταση, ούτε το πρόβλημα. Μας είπανε για την κινητικότητα. Κινητικότητα, τι σημαίνει αυτό. Ε, αυτό είναι ε, μετανάστευση, αποδημία, εξορία διαρροή εγκεφάλων. Φεύγουν χιλιάδες νέοι. Ό,τι έχουμε επενδύσει για να έχουμε νέους μορφωμένους για το μέλλον της χώρας μας, το χάνουμε. Σηκώνονται και φεύγουν. Δεν έχουν προοπτική στη χώρα. Σε λίγα χρόνια ποιος θα πληρώνει την κοινωνική ασφάλιση. Ποιος θα διατηρεί το κράτος. Ποιος θα διατηρεί τις κοινωνικές υπηρεσίες όταν φεύγουν οι νέοι και τις δημόσιες υπηρεσίες. Άλλη λύση, η πρωτοβουλία για την ε, ανεργία των νέων. Ούτε το 5% δεν δώσανε από αυτό που χρειάζεται είναι τεράστια τα προβλήματα για τις φτωχές χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις επιδοτούνται ασκήσεις, στάζ ή επισφαλής ε, θέσεις εργασίας. Ε, τι γίνεται με τους νέους. Δεν είναι αρκετά απασχολήσιμοι, δεν είναι αρκετά ε, καταρτισμένοι. Είναι καταρτισμένοι. Βελτίωση χωράει. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Πρέπει να έχουμε πολιτικές που να δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, να φτιάχνουν δουλειές, κοινωνική ανάπτυξη, πρόοδος, ε, συντονισμένη ε, βορρά-νότου και να μην βυθίζουμε στη λιτότητα και στις περικοπές των νότων, να το βοηθήσουμε να, βγάλει, να σηκώσει κεφάλι θα πρέπει να σκεφτούμε αυτές τις πολιτικές για μια νέα βιομηχανία σε τομείς που δημιουργούν ευκαιρίες, όπως είναι η πράσινη οικονομία, η ενεργειακή μετάβαση και να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες στην Ευρώπη. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε δουλειές και θα προστατεύσουμε την παραγωγή μας, τα εργοστάσια μας, τη βιομηχανία που τα ξεπουλάμε με τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και την άρση κάθε οικονομικού και εμπορικού φραγμού. Ευχαριστώ. Η Μαρ Αγγούλο από την Ισπανία και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένη ότι η απασχόληση είναι καλύτερη δυνατή κοινωνική πολιτική. Η εμπειρία της Ισπανίας και το μεγάλο δίδαγμα είναι αυτό που βγάλαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το ξέρουμε ότι δεν νοείται κοινωνική πολιτική αν δεν υπάρχει σωστή ε, κατεύθυνση και διακυβέρνηση της οικονομικής πολιτικής και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ε, η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην εξυγίανση του προϋπολογισμού. Γίνεται μια συζήτηση αν η λιτότητα ε, στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Στη χώρα μας υπήρχαν πολλά ελλείμματα. Τα ελλείμματα ήταν εκείνα που στραγγάλιζαν και έπνιγαν την ανάπτυξη. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και η εξυγίανση του προπολογισμού ήταν ο πρώτος πυλώνας που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να ξεφύγουμε από την ύφεση και να μπούμε στην ανάπτυξη και να σταματήσει η καταστροφή και αποδόμηση θέσεων εργασίας και να δημιουργηθούν νέες. Οι επενδύσεις είναι πιο κοινωνικές όσο δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Στην Ισπανία υπάρχει και ένας δεύτερος πυλώνας του κοινωνικού κράτους που είναι οι ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Από την αγορά εργασίας ξεκινήσαμε και στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Και μάλιστα ενώ είχαμε χαμηλή ανάπτυξη, σχεδόν 1%, λίγο παραπάνω, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας και πέρυσι μάλιστα 678.000. 14% συμβάσεις αορίστου χρόνου αυξήθηκαν. Σημαντικά μέτρα όπως είναι τα μέτρα εκείνα που ε, καταπολεμούν την ανεργία των νέων. Δεν χρειάζεται εδώ καμία συγκατάβαση ή αυταρέσκεια, αλλά όντως ήταν, άγγιζε το 50% η ανεργία των νέων, αλλά είχαμε φτάσει μέχρι και στο 55%. Άρα έχουμε 10% μείωση ήδη. Τέλος, Πρόεδρε, το κοινωνικό μοντέλο είναι Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες των κρατών μελών, αλλά και η ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επανέλθουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, και η εγγύηση για την νεολαία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Προτελευταίος ο Βλαντιμίρ Μαρίνκοβιτ από τη Σερβία. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση παρότι δεν είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόσουμε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μου και έχουμε πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έχουμε προσελκύσει κάποιους μεγάλους επενδυτές τα τελευταία χρόνια από τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Συνεχίζουμε να έχουμε σημαντικό πρόβλημα ανεργίας των νέων, η οποία ξεπερνάει το 40% στην ε, Σερβία. Αυτό βέβαια ισχύει και για το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων. Για το λόγο αυτό ε, η κυβέρνηση το 2016 το ε, προκήρυξε έτος της επιχειρηματικότητας. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την κυρία Βαντερμπουρκ και έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιονομικά κίνητρα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στις κάτω χώρες. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης ε, αυτών των επιχειρήσεων ε, στις κάτω χώρες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο τελευταίος ηλικιώτης, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι από μόνη τη η αλλαγή ρητορική και προσεγγίσεων τη Επιτροπή δείχνει τη χειροτρεύση τη κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία. Και η άποψή μα είναι ότι αυτή η χειροτρεύση οφείλεται κυρίω λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τη σκληρή λιτότητα, την πρόθεση του καπιταλισμού καζίνο, του οικονομικού συντονισμού από τι Βρυξέλλε, γιατί γίνεται με έναν τρόπο παράδοξο, αλλά και από την απορρίθμιση τη αγορά εργασία λόγω και όλων των πιο πάνω. Το μεγαλύτερο βάρο τη απορρίθμιση τη αστάθεια, τη επισφάλεια και τη φτώχεια το επομίζεται η νέα γενιά και οι ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού. Η νεανική ανεργία βρίσκεται στα πιο ψηλά επίπεδα που βρισκόταν στην ιστορία τη Ένωση. Η γενική ανεργία δε στι χώρε του Νότου ανέβηκε σε επίπεδα ρεκόρ. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα, διότι το ακούσαμε πολλέ φορέ από την Επιτροπή. Όταν έχουμε κριτήρια οικονομίστικα, οικονομικά, για το σύμφωνο σταθερότητα, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, γιατί δεν έχουμε και κριτήρια για το ποσοστό ανεργία, για το ποσοστό ανεργία των νέων, ε, όταν κρίνουμε τι οικονομίε στον χώρο. Γίνεται από όλου παραδεκτό πω η δημιουργία νέων θέσεων εργασία πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά για να γίνει αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα από το πολυδιαφημισμένο σχέδιο Γιούνκερ αφού πρόκειται κατά την άποψή μας για φρούδες ελπίδες ότι από μόνο το ιδιωτικό τομέα μπορεί να κινήσει την οικονομία. Γιατί το λέω αυτό. Από τα 315 δισεκατομμύρια του πακέτου Juncker, τα 295 δισεκατομμύρια πρέπει να τα επενδύσει ο ιδιωτικό τομέα. Ενώ αρχικά το σχέδιο Juncker, οι σκέψει του Juncker, όταν ήταν υποψήφιο, ήταν διαφορετικά. Και ξέρετε, από τα 16 δισεκατομμύρια ε, που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι από περικοπές από άλλα κονδύλια. Έχουν περικόψει 3,3 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα Συνδιώντας την Ευρώπη. 2,7 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Άρα δεν μιλούμε για ε, φρέσκο χρήμα. Η δική μας άποψη είναι ότι για να δημιουργηθούν πραγματικά συνθήκε ε, και νέες εργασίας αξιοπρεπής Χρειάζεται να προωθηθούν δημόσιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω της στήριξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ε, για να δημιουργηθούν ασφαλείς αξιοπρεπείς εργασίας, να αποτελούν μέρος μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης δημόσιας στρατηγικής, η οποία βεβαίως θα δημιουργεί και συνθήκες για ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλά το κράτος είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος επενδυτής και από το κράτος πρέπει να ξεκινούμε. Επίσης θα είναι μια στρατηγική η οποία πάνω απ' όλα θα σέβεται τις δημόσιες συμβάσεις, θα δυναμώνει τον κοινωνικό διάλογο και θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις μισθούς και κοινωνικές παροχές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε τις απαντήσεις των δύο μιλητών μας. Πόσο χρειάζεστε, ας πούμε πέντε λεπτά έκαστος και βλέπουμε για αρχή. Όπως θέλετε, με τη σειρά που θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, Άκουσα προσεκτικά την όλη συζήτηση. Αναφερθήκατε σε νέε θέσει απασχόληση και είπατε ότι αυτή είναι η πρωταρχική προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σαφέ. Από πού θα προκύψουν όμω αυτέ οι νέε θέσει απασχόληση. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι υπηρεσίε παροχή φροντίδα στου ηλικιωμένου, για παράδειγμα, ένα τομέα που μπορεί να δημιουργήσει νέε θέσει απασχόληση. Ορισμένοι αναφέρθηκαν σε άλλου τομεί βλέπουμε ότι όντως ο τομέας αυτός ε, παρουσιάζει αύξηση, ότι υπάρχουν νέες θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν εκεί. Στην ε, Τσεχία, στο παρελθόν, είχαμε ένα Συμβούλιο Ανάπτυξης ε, Ανθρωπίνων Πόρων. Τα συμβούλια αυτά είχαν περιφερειακό χαρακτήρα και ουσιαστικά προσπαθούσαν να προβλέψουν και να εκτιμήσουν τις ανάγκες απασχόλησης τα επόμενα πέντε χρόνια. Είχαμε προγράμματα επαγγελματικού επαναπρασαντολισμού, ή απόκτησης νέων δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενοι να αποκριθούν σε νέες θέσεις απασχόλησης που απαιτούν νέες δεξιότητες. Αλλά ακόμα και μετά από αυτή την επιμόρφωση δεν μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν θέσεις απασχόλησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα μια ευφυή προσέγγιση και να μπορούμε να κάνουμε και κάποιες προβλέψεις επομένως. Κάτι ακόμα που θέλω να θίξω. Η αδήλωτη εργασία ή η παρανομη εργαζόμενη. Ξέρετε ότι στην Τσεχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταβάλουμε έναν αγώνα κατά του φαινομένου αυτού και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας, έχουμε περισσότερους τέτοιους επιθεωρητές, έχουν περισσότερους πόρους οι άνθρωποι αυτοί, προκειμένου να πατάξουν αυτό το φαινόμενο των παράνομων εργαζομένων και της αδήλωτης εργασίας. Βέβαια δεν έχουμε το επίπεδο παρακολούθησης ή εποπτείας που έχουν άλλες χώρες όπως η Ισπανία. Επίσης αναφερθήκατε και σε άλλα ζητήματα όπως οι επενδύσεις στις υποδομές. Όσον αφορά την Τσεχία, θεωρώ ότι ε, οι επενδύσεις αυτές βρίσκονται σε καλό επίπεδο και μάλιστα παρέχουν πολλές νέες ευκαιρίες για νέες θέσεις απασχόλησης και σίγουρα οι επενδύσεις αυτές έχουν βοηθήσει να κρατήσουμε χαμηλά τα επίπεδα της ανεργίας. Ενδεχομένως να μην μπορούν όλες οι χώρες να εφαρμόσουν με τον ίδιο ποδοτικό τρόπο αυτές τις επενδύσεις, όπως δηλαδή έλαβαν χώρα στην Τσεχία, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι ε, οι επενδύσεις αυτές τις υποδομές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την ανεργία. Αν δεν καταφέρουμε μέσα σε δύο περίπου χρόνια να πετύχουμε το στόχο αυτό της μείωσης ανεργίας, καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί όλο και περισσότερο η δυσπιστία των εργαζομένων απέναντι στις κυβερνήσεις τους και απέναντι στο γενικότερο σύστημα το οποίο υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό με τη σειρά του μπορεί να τροφοδοτήσει περισσότερο τον πολιτικό εξτρεμισμό. Δύσκολο λοιπόν να βρει κανείς την κατάλληλη λύση, δύσκολο να καταλήξουμε σε ισορροπημένες λύσεις, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειώσουμε την ενέργεια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κυρία ευχαριστώ. Έχουμε διερμηνία, θα τα πω Ολλανδικά. Πρώτον, οι κάτω χώρες δεν είναι ένα κράτος όπου διακρίνεται για το διαλυμένο κοινωνικό κράτος. Έχουμε από τους υψηλότερους κατώτερους μισθούς και τα καλύτερα επιδόματα. Άρα εγώ τι λέω, μια αντιγωνιστική οικονομία θα πρέπει να έχει και μια ανθούσα επιχειρηματικότητα και ε, ένα καλό κοινωνικό κράτος. Και όποιος ισχυρίζεται ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν, εγώ το διαψεύδω, γιατί το ζω στη χώρα μου. Αυτό σημαίνει βέβαια ε, πάντα ε, μέτρα για να εξασφαλίζεις ότι είναι βιώσιμο το σύστημα. Την περασμένη περίοδο είχαμε και συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ολλανδία που δεν είναι εύκολο και είχαμε τους φιλελεύθερους ε, με τους σοσιαλιστές. Αυτοί οι δύο δεν είναι φυσικοί σύμμαχοι, είναι ένα δίπολο στο κοινοβούλιο, ένας απέναντι στον άλλον. Παρ' όλα αυτά κάνανε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στις συντάξεις και στην αγορά εργασίας. Οι μη φυσικοί σύμμαχοι. Ε, ευτυχώς, βέβαια και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν βουλευτές που αναλαμβάνουν δράση και δεν λένε μόνο στην Ευρώπη τι πρέπει να κάνει εκείνη, αρχίζουμε και έχουμε δράση σε εθνικό επίπεδο. Και δεν είναι ε, ε, εύκολη η καιρή, έχουμε πρόβλημα ανεργίας των νέων ε, και εκείνων που είναι ηλικία άνω των 50 ετών. Είναι χαμηλή βέβαια η ανεργία, σε εμά είναι 6%, αλλά όταν απολύονται εργαζόμενοι που είναι 50 και άνω δεν βρίσκουν δουλειά ή ε, όταν κλείνει η επιχείρησή τους. Ε, έχουμε και πολλούς αυτοπασχολούμενους. Αυτό είναι απάντηση στην ε, μη ευέλικτη αγορά εργασίας. Είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι αυτό που λέτε εδώ ότι χρειαζόμαστε ασφαλείς θέσεις διαβίου ορισμένη, αυτό είναι παλιά νοοτροπία. Θα πρέπει να έχουμε συστήματα που θα υποστηρίζουν τους ανθρώπους να πατάνε στα πόδια τους, να είναι και ευέλικτοι. Δηλαδή δεν έχεις μια δουλειά για πάντα. Μπορείς να αλλάζεις και δουλειά, μπορεί να αλλάζεις και επάγγελμα. Δεν σημαίνει ότι έχεις ε, απόλυτη ευελιξία και ανασφάλεια, αλλά ο κόσμος θα πρέπει να αποκτήσει εκείνη την ασφάλεια για να μπορεί να προσαρμόζεται σε νέες δουλειές. Και στην Ολλανδία αυτό δεν το έχουμε κατακτήσει, αλλά το δουλεύουμε. Γιατί χρειάζεται αυτό. Ας πούμε κάποιος ε, δουλεύει κάπου 10 χρόνια και μάλλον σε 10 χρόνια περίπου τα μισά επαγγέλματα και οι μισές θέσεις εργασίας δεν θα υπάρχουν. Σε 10 χρόνια ο μισός εργαζόμενος πληθυσμός θα δουλεύει σε τομείς που δεν τους έχουμε καν διανοηθεί ακόμα, που δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι θα είναι αυτά. Και πότε, πώς να έχεις λοιπόν μια θέση για όλη σου τη ζωή εκεί. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού, εξού και η παρέμβασή μου ότι υπάρχουν τελικά αυτοί που δημιουργούν τις θέσει δουλειά είναι οι επιχειρήσεις, όχι τα κρατικά όργανα. Κοστίζουν σε συνεργασία όμως πάντα με τις επιχειρήσεις και αυτές οι ευφύης πόλεις που είπαμε μπορούν να παίξουν ρόλο οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και να επενδύουν σε σχολεία, σε δρόμους κτλ. Γιατί ένας καλός πληθυσμός, καλά καταρτισμένος και μορφωσμένος είναι η βάση για το μέλλον. Έγινε μια ερώτηση, ψάχνω, ποιο το ρώτησε, ο συνάδελφο από τη Σερβία, για το καλύτερο τρόπο χρηματοδότηση των νεοφιών επιχειρήσεων. Εμείς τι έχουμε διαπιστώσει, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές αλλά και startups δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο. Και στο Υπουργείο Οικονομικών ε, της Ολλανδίας έχουμε μια διευκόλυνση έτσι ώστε να μπορούν να ε, κάνουμε καινοτομία και στρατηγική έρευνα ε, και αναλαμβάνει λίγο το κράτος χρηματοδότηση για να ε, χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι πάρα πολύ καχύποπτες και πολύ επιφυλακτικές μετά τη χρηματοοικονομική κρίση και τώρα τι θα κάνουμε. Ε, οι νεοφύης ψάχνουν νέο τρόπο χρηματοδότησης. Ένας τρόπος είναι το crowdfunding, άλλο είναι η επένδυση από άλλες επιχειρήσεις που επενδύουν σε νεοφύης και κάποιοι Άνθρωποι ε, λένε ότι σε 20 χρόνια από σήμερα οι τράπεζες δεν θα είναι ο υπαριθμόν ένα χρηματοδότης, θα έχουμε άλλες μορφές. Ε, άρα πρέπει να είμαστε στραμμένοι και προς το μέλλον και όχι προς το παρελθόν τι είχαμε, τι χάσαμε. Τι έχουμε στο μέλλον να κερδίσουμε. Και κάποιος από την Ιταλία είπε ότι δεν μπορούμε ως Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Μα έχουμε μια καταπληκτική αγορά, έχουμε, πώς να το πω, ε, ανθρώπους πολύ καταρτισμένους, μορφωμένους και ανθρώπινο δυναμικό ποιοτικό και ως Ευρωπαίοι έχουμε δώσει δείγματα γραφής τέτοια. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, για όλες τις χώρες, σε κάθε μια με τον τρόπο της, ότι ακριβώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Και όταν μιλάτε για τον ανταγωνισμό με την Κίνα, ναι είναι μεγάλος ανταγωνιστής, αλλά στην ε, Ολλανδία βλέπουμε ε, να επιστρέφουν πολλές δουλειές, γιατί εμείς είμαστε και πιο έξυπνοι και τα κάνουμε καλύτερο τρόπο από την Κίνα. Είναι πιο ποιοτικά τα προϊόντα και συνεργάζονται τα πανεπιστήμια και έχουν μια πολύ καλή θέση και κάνουν θεμελιώδη έρευνα ε, αλλά και προσαρμοσμένη. Και εκπαιδεύουν κόσμο που είναι για την πραγματική δουλειά, για την πραγματική αγορά εργασίας. Συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και είναι τεράστια δυναμική εκεί και είναι πολύ πιο παραγωγική από κάποιες άλλες αναντιστοιχίες που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και αυτό έχει να κάνει και με την κατάρτιση του, επαγγελματικού, του εργαζομένου πληθυσμού, γιατί όταν δεν είναι καλά καταρτισμένος τότε ε, βρίσκει δουλειά που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να την κερδίσουμε απέναντι στην Κίνα ως Ολλανδία ποτέ, δηλαδή ο πιο φτηνός. Γι' αυτό ποντάρουμε ε, στη μόρφωση του πληθυσμού και στις ψηλές και ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Αυτό συνεχώς χρειάζεται συντήρηση ε, δεν το έχουμε λύσει, αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα τα καταφέρουμε μαζί στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε και κάτι κοινό για να αγωνιστούμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η συζήτηση έδειξε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ε, στην ε, εκπαίδευση, την ε, ανάπτυξη, την έρευνα, την ενέργεια. Το πρόβλημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε αυτές. Η ιδέα του Juncker καταρχήν δεν είναι κακή ε, να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων. Το θέμα είναι όμως πώς θα χρηματοδοτηθεί. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με μεταφορά άλλων πόρων ε, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Θα πρέπει ε, να εισρεύσει φρέσκο χρήμα και θα πρέπει να συμμετάσχουν και ιδιωτικοί επενδυτές. θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις από τους ε, ανθρώπους με τα υψηλότερα εισοδήματα, για παράδειγμα. Ε, και νομίζω ότι μέχρι τώρα το σχέδιο Juncker υποχρηματοδοτείται και θα πρέπει και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο να σκεφτούμε πώς μπορούμε με αλληλεγγύη να πετύχουμε περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη για να δημιουργήσουμε ε, καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Ήταν ε, σωστή η παρατήρηση που έγινε. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα να μεταφέρουμε χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις χώρες που έχουν ε, πληγεί χειρότερα από την κρίση ώστε ε, να μην έχουν γραφειοκρατικά εμπόδια και να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση. Η Μπριγκίτε ε, με παρακινεί λίγο πολύ να περάσω στην τελευταία μου παρατήρηση ότι σε 30-40 χρόνια πολλές ε, θέσεις απασχόλησης ε, το 50% των θέσεων απασχόλησής μας δεν θα υπάρχει πια. Όταν ερευνητές και επιχειρηματίες μας λένε ότι έχουμε περάσει στην επόμενη βιομηχανική επανάσταση με την ψηφιοποίηση. Και μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 30 ή 40%. Ε, τότε αυτή η αύξηση είναι διπλάσια ε, στη Γερμανία σε σχέση με ε, τα προηγούμενα 40 χρόνια και ε, και έτσι δεν χρειάζεται πια να συζητάμε για τους στόχους της απασχόλησης ε, για μέχρι το 2020. Θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα που θα συμπληρώσουν το κενό, λένε κάποιοι. Ε, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει αυτόματος. Θα πρέπει να διαμορφωθεί σωστά η πολιτική και η οικονομική διαδικασία που θα μας φέρει εκεί. Δεν αρκεί να πούμε ότι εντάξει όλα είναι καλά, ούτε κατηγορώ κανένα να το κάνει αυτό, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τις εξελίξεις στο μέλλον και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ε, δώσουμε δουλειά στους ανθρώπους ε, από την οποία να μπορούν να ζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ε, Πυρκίτε Φαντενκούρκ και Γιάροσλαβ Τσάλατιλ, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Και κλείνω έτσι την συνεδρίαση. Θα τα πούμε απόψε στο γεύμα και στο δείπνο και αύριο στην συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ.